Ε, good afternoon, ladies and... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ, καθίστε. Θα ξεκινήσουμε σε ένα λεπτό. Έχουμε λοιπόν λίγο χρόνο για να καθίσουμε ο καθένας όσο πιο άνετα μπορεί και να ολοκληρώσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει. Uh, let me welcome. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους, κυρίως όμως την Επίτροπο και την υποδιορισμό και την uh, Αντιπρόεδρο για την Ενεργειακή Ένωση, την κυρία Αλένκα Μπρατούσεκ, η οποία είναι πρώην Πρωθυπουργό της Σλοβενίας. Η δημόσια αυτή ακρόαση έχει οργανωθεί από κοινού από τις Επιτροπές Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, τον συνάδελφο Τζοβάνι Λαβία Πρόεδρο και την και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Ήτρε, ε, ε, ε της οποίας εγώ είμαι ο πρόεδρος και βλέπετε εδώ μπροστά το όνομά μου, κύριος Μπούζεκ. Θα είμαστε και οι δύο συμπρόεδροι της ακρόασης αυτής. Επίσης θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην αίθουσα αυτή, τα μέλη των δύο επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και εκπροσώπους των ευρωπαϊκών εταιριών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ε, από τα κράτη-μέλη, όπως επίσης Πρέπει να πω ότι η δημόσια αυτή ακρόαση μεταδίδεται διαδικτυακά από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι λοιπόν οι Ευρωπαίοι που μας παρακολουθούν είναι και αυτοί ευπρόσδεκτοι. Θα ήθελα να πω ότι κάθε επιτροπή είναι εν γέννη υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή πολιτική ενέργεια, την ασφάλεια της ε, προμήθειας ενέργειας, την ε, εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προώθηση της διασύνδεσης των ενεργειακών αγωγών και τη δημιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών. Η ενεργειακή πολιτική θα είναι ένα σοβαρό θέμα στην νομοθετική μας εργασία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας να ακούσουμε από την κυρία Αντιπρόεδρο, την υποδιορισμό επίτροπο, πώς σκοπεύει να χειριστεί τις δυσκολίες αυτές. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ζητήματα όπως ο ανταγωνισμός, οι εξωτερικές σχέσεις, ή τα θέματα της βιομηχανίας μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης. Όλοι σας, αγαπητοί συνάδελφοι, και από τις δύο επιτροπές, και την ΕΝΒΙ και την Ήτρε, έχετε πάρει, έχετε λάβει όλα τα έγγραφα. Το, την επιστολή ανάθεση στην κυρία ε, Επίτροπο, το βιογραφικό της σημείωμα, την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και της Επιτροπής νομικών υποθέσεων, όπως επίσης και τις γραπτές απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Υπάρχει το ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις στις θέσεις Και βεβαίως, πριν δώσω το λόγο στο συνάδελφο για να προεδρεύσει και αυτός, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποδιορισμό επιτρόπους με βάση την, τις γενικές τους ικανότητες, την αφοσίωσή τους στην Ευρώπη και την προσωπική τους ανεξαρτησία. Επίσης, αξιολογεί τη γνώση του τομέα στον οποίο, τον οποίο θα αναλάβουν, όπως επίσης και τις δεξιότητές τους στον τομέα της επικοινωνίας. Ε, Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω την ε, υποδιορισμό επίτροπο και αντιπρόεδρο η υπεύθυνη για την Ενεργειακή Ένωση, την κυρία Λένκα Μπράτουσεκ αφού διαδραμάτισε αρκετούς ρόλους ε, στο εσωτερικό της ε, σλοβενικής κυβέρνησης, της σλοβενικής δημόσιας διοίκησης, ξεκίνησε την καριέρα της στο πολιτικό επίπεδο το 2011 ε, ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Σλοβενικού Κοινοβουλίου και το Φεβρουάριο του 2013 έγινε πρωθυπουργό της Σλοβενίας. Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό που ε, ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα. Το 2014 ανέλαβε και το Υπουργείο Υγείας. Ε, Στου τομεί της αρμοδιότητές της ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση του έργου διαφόρων επιτρόπων και κυρίως ε, του Επιτρόπου για την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια και του Επιτρέπου για το Περιβάλλον της θαλάσσιες πολιτικές και την αλληλεία που καλύπτουν μεγάλο τμήμα των καθηκόντων του Επιτρόπου για το Περιβάλλον θα πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική ενεργειακή ένωση με ε, σημαντικό ρόλο για την αλλαγή του κλίματος και θα πρέπει να καθοδηγήσει τις βασικές αρμοδιότητες και να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέτει και ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη της ε, ε, θέσεων εργασίας της πράσινης ανάπτυξης και θέλει να κάνει την Ευρώπη ε, ηγέτη στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Γι' αυτό και ακριβώς και το χαρτοφυλάκιό της είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την οποία προεδρεύω. Εδώ και πολλά χρόνια δίνουμε μάχη για μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση, μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και βιώσιμης είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ηγετικό ρόλο και πολύ καλά συντονισμένος Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες ε, παγκόσμιες διασκέψεις ε, για το κλίμα εν ώψη και διάσκεψη του των Παρισίων του 2015. Επίση, να υπάρχει και ε, κατάλληλη προοπτική για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και η ανάγκη φυσικά μεταρρύθμισης τη αγορά άνθρακα και το σύστημα ανταλλαγών εκπομπών, τα λεγόμενα ETS. Μετά από αυτά να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μπούζεκ για να μας εξηγήσει λίγο πώς ακριβώς ε, θα γίνει η ακρόαση. Σας ευχαριστώ συνάδελφε, σας ευχαριστώ και για τα εισαγωγικά σας σχόλια και να σας πω το εξής. Στην αρχή της ακρόασης η υποψήφια επίτροπος θα κάνει μια εναρκτήρια δήλωση και Στην περίπτωση των ακροάσεων της Επιτροπής Ήτρε είχαμε 15 λεπτά για την ε, ε, ομιλία, ενώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι 10 τα διαθέσιμα λεπτά. Συμφωνήσαμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην υποψήφια Επίτροπο για 12 λεπτά. Ε, ένα ενδιάμεσο, ένα μέσο όρος μεταξύ των δύο επιτροπών. Ενημερώθηκε η υποψήφια Επίτροπος για την απόφασή μας, επομένως θα μιλήσει για 12 λεπτά. Αυτά στην αρχή. Στη συνέχεια, στο τέλος της ακρόασης θα της δοθούν 5 λεπτά για τις ε, καταλεκτικές ε, ε, παρατηρήσεις της. Από εκεί και πέρα, ό συνήθως, θα έχουμε 45 λεπτά, 3 λεπτά για την κάθε ερώτηση, 1 λεπτό για την ερώτηση και 2 λεπτά για την απάντηση. Επίσης, να σας πω ότι για όλους τους συναδέλφους ισχύει αυτό και για την προτινόμενη επίτροπο, θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης. Θα υπάρχουν 5 δευτερόλεπτα επιπλέον ανοχής για τους συναδέλφους και 10 δευτερόλεπτα για την υποψήφια επίτροπο και από εκεί και πέρα θα κλείνει το μικρόφωνο. Ορισμένε φορέ δεν είμαστε τόσο αγενεί, αλλά σε γενικέ γραμμέ έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Επομένω, είναι στο χέρι μας πριν ε, λήξει ο χρόνος, 10 δευτερόλεπτα πριν, θα αρχίσει να ανάβει ένα, ε, δύο αστεράκια στο τραπέζι. Επομένως, ε, κύριε Προτινόμενη Επίτροπε, θα δείτε ότι θα αναβοσβήνουν αυτά τα αστεράκια για να ξέρετε ότι ολοκληρώνεται ο χρόνος σας. Ο πρώτος γύρος ερωτήσεων θα είναι από εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Υπάρχει διερμηνία σε 23 γλώσσες, επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μητρική σας γλώσσα. Σας παρακαλώ να μην μιλάτε πολύ γρήγορα, διότι πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διερμηνία. Η ε, συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορείτε να έχετε και πρόσβαση σε μαγνητοσκόπηση της ακρόασης ε, στην ίδια ιστοσελίδα. Ήγηκε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσει η ακρόαση μετά από όλες αυτές τις αρχικές παρατηρήσεις. Ε, Κύρια Επίτροπη Υποδιορισμό, τέος Πρωθυπουργέ, να σας δώσω το λόγο λοιπόν για να κάνετε τις αρχικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Ενώπιόν μας Έχουμε πέντε πολύ απαιτητικά χρόνια για τα οποία είμαι πεπισμένη ότι θα είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση είχε καταστροφικέ συνέπειε σε πολλές χώρες. Η ανεργία των νέων έχει φτάσει σε απαράδεκτα επίπεδα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τι ανάγκε των λαών τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι κρίσιμα στην αποκατάσταση εμπιστοσύνης απέναντι σε αυτό το θεσμικό όργανο. Γι' αυτό έχουμε ε, πρέπει να κάνουμε το θεματολόγιο για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή να επιτύχει. Αυτό το θεματολόγιο θα εφαρμοστεί από μια ισχυρή ομάδα μέσω αμοιβαία συνεργασία. Σε αυτή την αμοιβαία συνεργασία βλέπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως έναν από τους εταίρους κλειδί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να δεσμευτώ ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να ενισχύσω τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Ως πρώην Πρωθυπουργό και μέλος του Κοινοβουλίου βεβαίως εκτιμώ τη σημασία του συνεισφοράς του Κοινοβουλίου στην εξέβρεση λύσεων και βεβαίως την υλοποίηση της κοινή ατζέντα για προς των Ευρωπαίων πολιτών. Λοιπόν, αγαπητά μέλη, είναι τιμή για μένα και έρχομαι με μεγάλη ταπεινοφροσύνη για να καθίσω ενώπιόν σας ε, ω υποψήφια για τη θέση τη Αντιπροέδρου για την Ενεργειακή Ένωση. Η πατρίδα μου η Σλοβενία εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια πριν από 10 χρόνια. Για μένα αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Εγώ και η γενιά μου γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο χώρος στον οποίο ανήκουμε. Αποτελεί λύση, δεν είναι πρόβλημα. Και η δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης με την σύγκληση των κρατών μελών στον τομέα της ενέργειας και των πολιτικών για το κλίμα έχει κάθε δυνατότητα να αποτελέσει ε, έναν ένα βήμα προς την στρατηγική της Ευρώπης για να ξεπεραστεί η κρίση. Αυτό ακριβώς είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ όταν απευθύνθηκε στο Κοινοβούλιο και αυτό είναι και το όραμά μου. Η εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά και η ενίσχυση μιας βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης με βάση ξεκάθαρους στόχους για το κλίμα, όπως επίσης ε, ε, και άλλοι, άλλοι στόχοι που αποτελούν τις βασικές προκλήσεις της εποχής μας. Ως μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που μέχρι πρόσφατα, έχω πλήρη συνέστηση το πόσο σύνθετα είναι τα θέματα της ενέργειας. Όχι μόνο έπαιξα ενεργό ρόλο ε, στη στρατηγική των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ήμουν απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, είμαι περήφανη να πω ότι κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργία μου στη Σλοβενία μπορέσαμε να υλοποιήσουμε το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Κυρίες και κύριοι, ε, ανέλαβα πρωθυπουργό σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία του νεαρού μας κράτου και ε, πραγματικά μέσω μιας σωστά μετρημένης και συνεπούς πολιτικής με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές και τις δεσμεύσεις μας καταφέραμε να βγάλουμε τη Σλοβενία από την χειρότερη οικονομική κρίση. Πιστέψτε με, είμαι συνηθισμένη να δουλεύω σε συνθήκες υψηλού στρες, επίσης όμως γνωρίζω ότι το άγγιγμα της γυναίκας καμιά φορά μπορεί να ερεμεί στα πράγματα. Θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια για τον ορισμό μου ως επιτρόπο. Όπως θα γνωρίζετε ε, υπήρχε μια προθεσμία υποβολή των ονομάτων των υποψηφίων και αυτή ήταν το τέλος Ιουλίου. Δεδομένου ότι δεν μπορούσε να επιτεθεί συμφωνία ανάμεσα στους εταίρου του συνασπισμού ε, και δεν υπήρχε ένας ε, υποψήφιος, είχαμε δύο δυνατότητες. Είτε να μην στείλουμε κανένα όνομα στις Βρυξέλλες και να περιμένουμε τη νέα κυβέρνηση να το κάνει στο τέλο Σεπτεμβρίου και όλοι φαντάζεστε τι επιπτώσει θα είχε αυτό στην Επιτροπή ή να στείλουμε έναν κατάλογο ονομάτων. Αυτός ο κατάλογος το από τρία ονόματα, συμπεριλαμβανομένη και του δικού μου και την τελική απόφαση την έλαβε ο πρόεδρος Γιούγκερ. Αυτά συνέβησαν και τίποτε άλλο. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στην κοινή μας πρόκληση, τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης. Η πατρίδα μου δεν είναι η μόνη χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λόγω της γεωγραφικής της θέσης ε, ε, αντιμετωπίζει κινδύνους στην ενεργειακή ασφάλεια όπως μια, την υπερβολική εξάρτηση από έναν μη Ευρω... κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης προμηθευτή. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να, με... να πιστώ ότι κανένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές δυσκολίες από μόνος του. Οι ενεργειακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν απαιτούν τώρα περισσότερο από ποτέ μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη που θα μιλάμε μια φωνή διεθνώς και, ένα καλά, και μια καλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει 53% της ενέργειάς της. Αυτά τα νούμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να καταλάβουμε τη σημασία του έργου της ε, ε, Ενεργειακής Ένωσης. Καθημερινά εισάγουμε ενέργεια αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το 2013 το κόστος της ενέργειας έφτασε 400 δισεκατομμύρια ευρώ και ήταν το 1 πέμπτο του συνόλου των εισαγωγών μας. Η εξάρτηση από τις εισαγωγές από μόνη της αποτελεί κίνδυνο, αλλά όταν αυτό συνδυάζεται με εξάρτηση από έναν μοναδικό εταίρο, τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν. Το γεγονός ότι έξι κράτη-μέλη ε, στηρίζονται αποκλειστικά σε, ένα, σε μια ξένη πηγή για την προμήθεια αερίου, ενώ πολλά άλλα έχουν έκθεση που ξεπερνά το 60% είναι γεγονός. Τα νούμερα αυτά μας δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το όραμά μας. Το όραμα μιας ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα συμπτύξουν μια ανθεκτική ε, ενεργειακή ένωση το όραμά μου είναι μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση η οποία θα, έχει, θα βλέπει στο μέλλον σε, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και η οποία θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και αύξηση της ασφάλειας ε, της, ενέργεια, της προμήθειας ενέργειας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και με την ε, διασύνδεση της ε, υποδομής με τους συνδετήριους αγωγούς, όπως επίσης και μια ενωμένη παρουσία στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Δεύτερον, να συνεχίσουμε να προωθούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διευρύνοντας την, ε, και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή κυριαρχία στην τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη μέσω πρωτοβουλειών ε, για τις επενδύσεις, την προώθηση της ε, ευαισθητοποίησης. Τρίτον, η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης ανάπτυξης με τη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την επίτευξη των στόχων του 2020 και, την, και τους φιλόδοξους στόχους για το 2030 ε, σε σχέση με τα κίνητρα που θα μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση και θα αυξήσουν την αποδοτικότητα της ενέργειας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η όπως βλέπουμε τα πράγματα σήμερα μπορεί να μοιάζει ότι η σχέση μας με τη Ρωσία είναι το κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, βραχυπρόθεσμα, η ασφάλεια της προμήθειας αερίου οπωσδήποτε είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την Ευρώπη και τους πολίτες στον τομέα της ενέργειας. Η επίτευξη των κλιματικών στόχων μας, ενώ ταυτόχρονα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πρέπει να παραμείνει πρώτη προτεραιότητα της ατζέντα μας. Είμαι πεπισμένη ότι ε, αν κάνουμε την, την εσωτερική ενεργειακή αγορά μία πραγματικότητα χωρίς επιστροφή και αν ε, εφαρμόσουμε τις, ε, τους κλιματικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί ξεκινώντας από το πακέτο 2020 σε συνδυασμό με ένα μεγάλο πακέτο επενδύσεων, εκτεταμένων επενδύσεων όπως ανακοίνωσε ο κύριος Γιούνκερ θα έχουμε το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε σωστά και την οικονομική και την κλιματική αλλαγή και τις δυσκολίες της εποχής μας. Μόνο επίσπευση των επενδύσεων στην ενεργειακή υποδομή, καθαρές ε, τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και κυρίως δοτική χρήση της ενέργειας μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Ε, το ενεργειακό πλαίσιο του 2030 πρέπει να μας καθοδηγεί. Κυρίες και κύριοι, αυτό φυσικά θα απαιτήσει και χρόνο και σκληρή δουλειά και απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι απολύτως προσιλωμένη στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τις Επιτροπές Ήτρε και Ένβη. Θα ήθελα να αναλύσουμε τις αλλαγές, τις δυσκολίες από κοινού, να αποφασίσουμε για συγκεκριμένες δράσεις και τις φιλοδοξίες για την εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης και τους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Αυτό θα μας ε, θα φέρει την αλλαγή. Η αλλαγή που χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη, νέε θέσει εργασία, ενώ θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργεια και θα ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια. Στο παρελθόν η Ευρώπη έχει δείξει ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη και μείωση τη κατανάλωση ενέργεια ταυτόχρονα. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερα και να το γνωρίζουν αυτό και οι πολίτε μα. Εάν θεωρήσουμε ότι το 50% τη ενέργεια ενέργειας χρησιμοποιείται για θέρμανση ψήξη, είναι προφανές ότι η δυνατότητα για εξοικονόμηση δεν έχει εξαντληθεί. Εδώ μπορούμε να πετύχουμε ταυτόχρονα δύο πράγματα. Η, ανανέωση, ενεργειακή ανανέωση των κτηρίων με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα, η θα μειώνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές. Αυτό είναι ένα είδος βιώσιμης ανάπτυξης που χρειάζεται η Ευρώπη. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε ένα σημαντικό κομμάτι των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα επενδυθούν και τα οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην εναρκτήρια ομιλία του να δοθεί προς έργα ενεργειακής απόδοσης που θα ενισχύσουν την πράσινη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο σωστός δρόμος για την Ευρώπη. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα απαιτήσει πραγματικά ομαδική δουλειά και συγκέντρωση ε, σε συγκεκριμένα έργα μεγάλης σημασίας. Επίσης από την πλευρά της Επιτροπής ε, στο πλαίσιο της, του θεματολογίου για τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή θα αναλάβω ενεργό ρόλο για τις δύο ε, βασικές προτεραιότητες. Θα συντονίσω και θα καθοδηγήσω τη δουλειά με τους ε, συναδέλφους επιτρόπους που, ε, αφορούν και που έχουν σχέση με την Ενεργειακή Ένωση. Θα είναι ε, καθήκον μου να εξασφαλίσω ότι οι ιδέες και λύσεις από, τη, από τους συγκεκριμένους τομείς να ενσωματωθούν στρατηγικά σε μια πραγματικά καλά συντονισμένη δράση. Μία ακόμα πρόταση αν αγαπητά μέλη της των Επιτροπών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, είπε η κυρία κλείνοντας την ομιλία της. Ευχαριστώ πολύ. Θα έλθουμε τώρα στις, στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και θα αρχίσουμε με τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Κάρινς. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπράτουσεκ, λέτε, αλλά θα κάνετε. Όταν κάποιο το σπίτι καίγεται, οι γείτονε τρέχουν να βοηθήσουν. Και αυτός που καίγεται το σπίτι του, πολύ ευχάριστα δέχεται τη βοήθεια. Όμως, όταν τα οικονομικά της χώρας σας ήταν σε μεγάλη δυσκολία, ως Πρωθυπουργός αρνηθήκατε την βοήθεια των Ευρωπαίων γειτόνων σας. Ερώτηση, αρνηθήκατε την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σύνθημα ότι η Ευρώπη δεν θα έλθει σε κατοχή της Σλοβενίας. Η ερώτησή μου είναι πώς θα δημιουργήσετε ενεργειακή ένωση, πώς θα σας εμπιστευτούμε να φτιάξετε την ενεργειακή ένωση, όταν λάβουμε υπόψη ότι με κάποιον τρόπο θα φάει αυτή η ένωση κάποια κάποιο κομμάτι από την ανεξαρτησία σας, όπως το καταλαβαίνετε εσείς τουλάχιστον, όπως το είπατε. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κυρία Ευρωβουλευτά. Είμαι πεπισμένη ότι είναι σωστό που υπάρχει μηχανισμός στήριξης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες που τον χρειάζονται. Ωστόσο είμαι υπερήφανη που η Σλοβενία μπόρεσε να λύσει τα προβλήματα μόνη της. Εγώ θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι η Σλοβενία αντίθετα με τις προσδοκίες πολλών δεν χρειάστηκε την βοήθεια αυτή, τη στήριξη αυτή. Καταφέραμε με κοινή προσπάθεια οι Σλοβαίνοι να δείξουμε στην Ευρώπη ότι δεν πέφτουν όλες οι χώρες όπως το ντόμινο, όπως ε, οι ψηφίδες του ντόμινο, αλλά ότι μπορούν να σταθούν και μόνες τους. Δεν απορρίψαμε την βοήθεια αυτή, τη στήριξη, καταφέραμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας και γι' αυτό είμαι ακόμη και σήμερα υπερήφανη. Τώρα η Ενεργειακή, η Ενεργειακή Ένωση αποτελεί ένα από τα κύρια καθήκοντα για την επόμενη πενταετία. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι θα είναι απαραίτητο η συνεργασία να είναι εντατική. Έχουμε βάλει κοινό στόχο να στήσουμε στα πόδια της μια ενεργειακή ένωση. Και γι' αυτό είναι σημαντικό οι χώρες μέλη να συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή, προς την επίτευξη των κοινών στόχων. Και βέβαια θα χρειαστούμε την βοήθεια όλων και την δική σας. Μόνη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μόνη μου εγώ ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους. Σε συνεργασία με εσά, με τις χώρες μέλη, σίγουρα ο στόχος αυτός είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Βαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε η έννοια της Ενεργειακής Ένωσης είναι ακόμα αρκετά ασαφής και θα έχετε και άλλες ερωτήσεις σχετικά. Ποια όμως είναι η συγκεκριμένη σχέση που θα έχετε εσείς ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την Ενεργειακή Ένωση και ο αρμόδιος για ενέργεια και κλίμα επίτροπος. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δυο σας και αν υπάρχει διαφορά και αν δεν υπάρχει διαφορά τι θα κάνετε ακριβώς. Για να καταστήσω σαφέστερη την ερώτησή μου, θα προσπαθήσω να διευκρινίσω λίγο περισσότερο. Ποιο θα είναι αρμόδιο, για παράδειγμα, για να θέσει του στόχου τη ενεργειακή αποδοτικότητα καθώ και του στόχου για τι ανανεώσιμε ενέργειε. Θα είναι ο Επίτροπος ενέργεια και κλίματο η Αντιπρόεδρος για την Ενεργειακή Ένωση. Και αν θα είστε εσεί, τότε ποιοι θα είναι οι στόχοι σα για την αποδοτικότητα τη ενέργεια. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Η απάντηση παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ευρωβουλευτά. Γνωρίζω ότι πολλούς απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθούν οι εργασίες της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι πεπισμένη ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ μελέτησε το θέμα πριν να κάνει τη σχετική πρόταση. Είμαι πεπισμένη ότι με την εργασία μας θα μπορέσουμε να πείσουμε ότι η Επιτροπή μας εργάζεται αποτελεσματικά. Εγώ θα συντονίζω και θα καθοδηγώ τις εργασίες πλειώνων επιτρόπων με ένα κοινό στόχο, τον συνδυασμό των στόχων των επιμέρους χαρτοφυλακίων, έτσι ώστε να συναποτελέσουν ένα ενιαίο στόχο. Είμαι πεπισμένη ότι θα τα καταφέρουμε, ότι θα συμφωνήσουμε βεβαίως με την προϋπόθεση ότι θα μας χορηγήσετε και εσείς την υποστήριξή σας, ότι θα καταφέρουμε να συνεννοηθούμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα μπορέσουμε να φέρουμε σε αίσιο πέρα στην αποστολή μας. Όσον αφορά τους στόχους και τις ευθύνες, τις αρμοδιότητες για την επίτευξή τους, Πιο σημαντικό είναι το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, αν θα μπορέσουμε να θέσουμε φιλόδοξους στόχους και αν θα συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους αυτούς. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρομαι συλλογικό στην ευθύνη για την επίτευξη των κοινών στόχων. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Γιάκεβιτς, εκ μέρους των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύρια Υποψήφια Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Επομένως, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα πρώτων υλών, η ασφάλεια εφοδιασμού, κυρίως ε, εξανατολών και η παρούσα κατάσταση μας υποχρεώνει να δράσουμε ταχύτατα για να υπάρχει ενεργειακή αποδοτικότητα. Η ασφάλεια εφοδιασμού ε, παρόλα αυτά εξαρτάται και από τη Ρωσία. Και όπως είπατε κι εσείς, Μας είπατε ότι είστε διατεθειμένοι να μας δώσετε ένα πρόγραμμα δράσης ε, ε, και υπάρχει και ο κανονισμός ε, για την ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί ταχύτατα. Εάν η Ρασία σταματήσει να παρέχει ανέργεια στην Ευρώπη, ποιος θεωρείτε ότι θα πρέπει να την αντικαταστήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμη Ευρωβουλευτή, όντως η ασφάλεια εφοδιασμού είναι ακρογωνίος λίθος της Ενεργειακής Ένωσης. Και λόγω της παρούσας κατάστασης είμαστε υποχρεωμένοι να δρούμε ταχύτατα. Έχουν υπάρξει στην, στο παρελθόν στην Ευρώπη κρίσεις ε, φυσικού αερίου και δύσκολα μπορεί κανείς να πει ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ε, η τελευταία κρίση, η πιο πρόσφατη άλλωστε, ήταν το 2009. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και βραχυπρόθεσμες λύθεις αλλά και μακροπρόθεσμες λύθεις. Βραχυπρόθεσμες με μια πιο ισχυρή αγορά, με καλύτερα διασυνδεδεμένες δομές και με καλύτερη μετάδοση ενέργειας μεταξύ των διαφόρων χωρών, μεταξύ των διαφόρων περιβεριών ε, και ε, μεταξύ των διαφόρων περιοχών μιας χώρας, ε, περιοχές που σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ακόμα διασυνδεδεμένες. Με άλλα λόγια, καλύτερες υποδομές. Αυτό θεωρώ ότι είναι θεμελιώδου σημασίας για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού. Τώρα, βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης σε επίπεδο διεύθυνσης υπάρχει ήδη κάτι τέτοιο, γίνονται κάποια τεστ αντοχής σε περίπτωση που μειωθεί για παράδειγμα ε, η ποσότητα φυσικού αερίου ή και διακοπεί πλήρως ε, ο εφοδιασμός σε φυσικό αέριο. Ε, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και φυσικά θα ε, δούμε και τι γίνεται από πλευράς Μεσογείου, Νορβηγίας. Ε, θα έχουμε στη διάθεσή μας και άλλους ε, προμηθευτές. Ευχαριστώ ο κύριος Φέντερλαϊ από πλευράς Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Κύρια Προτινόμενη Επίτροπε για την προκαταρκτική σας ομιλία η κλιματική αλλαγή και η παρούσα γεωπολιτική ε, κατάσταση μας έχει σφαίρει σε ένα στεαδροδρόμι από πλευράς Ευρώπης, είτε το επιθυμούμε είτε όχι. Οι θέσει εργασίας ε, και η ε, σταθερότητα εξαρτώνται από τη Ρωσία και από μια ταραγμένη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κατάλληλα μεταρρύθμιση ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να μειώσουμε και τις επιδοτήσεις σε αυτούς τους δικτάτορες. Η ερώτησή μου λοιπόν σε εσά, κυρία Υποψήφια Επίτροπε, είναι πώς θα διασφαλίσετε ότι οι επίτροποι για τους οποίους θα είστε αρμόδια θα ε, φροντίσουν να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε εναλλακτικέ πηγές ενέργειας η Ευρώπη. Ευχαριστώ η απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Το όραμά μας είναι σαφές. Οι στόχοι μας είναι σαφείς και ε, φυσικά και το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι σαφές. Θεωρώ ακράδαντα ότι αυτοί είναι κοινοί στόχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς τη βοήθεια των κρατών μελών, δεν θα μπορέσει να επιτύχει και πάρα πολλά στον τομέα αυτό. Επομένως, χρειάζεται συνεργασία και ε, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι όντως πρόκειται για κοινού στόχους. Επίσης να σας πω ότι χωρίς την ε, ε, συνδρομή των κρατών μελών και τη σύμφωνη γνώμη τους και χωρίς τη βοήθεια τη δική σας, εγώ δεν θα μπορέσω να αποδείχω και πάρα πολλά. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε όλοι για τον ίδιο κοινό στόχο. Ε, σκοπό. Οι εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια είναι πολύ σημαντικέ κατά την άποψή μου, διότι καταρχά μειώνουν τι εκπομπέ ε, των αέριων του φαινομένου θερμοκηπίου, αυτό είναι ο πρώτο βασικό στόχο, μειώνουν την εξάρτησή μα από εισαγωγέ και κάτι εξίσου σημαντικό, δημιουργούν νέε θέσει εργασία, τι λεγόμενε πράσινε θέσει εργασία Καθώ επίση ενισχύουν και την οικονομική μα ανάπτυξη. Βεβαίω, είναι σαφές για μένα ότι και βάσει της νομοθεσίας, βάσει των συνθηκών, τα κράτη-μέλη ανεξάρτητα ε, το καθένα είναι αυτά που αποφασίζουν για το ενεργειακό μείγμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουν στην επικράτειά τους. Παρ' όλα αυτά, ε, όλοι εμείς από κοινού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε κοινούς στόχους και θα πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι κοινοί στόχοι. Αν παρ' όλα αυτά θέλουμε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να είναι φθηνότερες, και να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση για τη βιομηχανία σε αυτές τις πηγές, τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας σε έρευνα και ανάπτυξη, γεγονός το οποίο σίγουρα θα μας βοηθήσει. Οι δικές μου προσπάθειες σίγουρα θα προσανατολιστούν προς μια Ευρώπη που θα έχει τα ενία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιλικιώτης, εξ ονόματος της Αριστεράς. Στην ανακοίνωση τη Κομισιόν τον περασμένο Μάιο με θέμα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αναφορά στα μεγάλα κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο ούτε στο πώ μπορούν να αξιοποιηθούν. Υπάρχει μόνο μια γενική αναφορά στη δημιουργία Μεσογειακού κόμβου ενώ ο πολύ σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο για την ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια τη Ένωση υποτιμάται. Πώ αντιλαμβάνεστε εσεί το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η περιοχή και ειδικότερα η Κύπρο, τη οποία η ΑΟΣ είναι πλούσια σε κοιτάσματα φυσικού αερίου. Είναι στι προτεραιότητε σα η ανάπτυξη ενό συγκεκριμένου σχεδίου δράση για την υλοποίηση ενό μεσογειακού κόμβου μέσω αγωγού προ την Ευρώπη. Σε ποιε ενέργειε θα προβείτε για την ανάπτυξη συνεργασιών με τι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Χθε η Τουρκία, μια υποψήφια προσένταξη χώρα, έχει προχωρήσει παράνομα στη δέσμευση περιοχών νοδιό τη Κύπρου, ε, ε, επηρεάζοντα τα κυριαρχικά δικαιώματα τη Κυπριακή Δημοκρατία και τη εταιρεία ΕΝΗ που δραστηριοποιείται σε αυτήν την περιοχή αυτή την περίοδο. Έληξε ο χρόνο σα. Παρακαλώ απαντήστε. Ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτά για την ερώτηση. Δεν είναι απαραίτητο νομίζω να τονιστεί ότι η ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας αποτελεί θεμέλιο της Ενεργειακής Ένωσης στην οποία προσβλέπουμε η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών θα είναι ένας από τους τρόπους να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους, έτσι ώστε η Ευρώπη να γίνει ενεργειακά πιο ανεξάρτητοι. Βέβαια ορισμένα βήματα πρέπει να ληφθούν ταχύτερα από άλλα. Όπου για άλλα θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Είναι γεγονός ότι ορισμένα έργα έχουν ήδη σχεδιαστεί και είναι πιο προχωρημένα, άλλα έργα χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Μια ισχυρή ενή αγορά είναι αυτό που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η Ενεργειακή Ένωση, ώστε η οικονομία μας να γίνει ανταγωνιστικότερη. Αν θέλουμε ωστόσο να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι, και είμαι πεισμένη ότι αυτός είναι ένας κοινό μας στόχος, όπως εξήγησα και πριν, τότε θεωρώ ότι πρέπει απαραίτητα να διαφοροποιήσουμε και τις ενεργειακές πηγές και τις διαδρομές της ενέργειας, όπως είπατε και εσείς. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μέσα στους επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστώ. Κύριε Τούρμες, εξ ονόματος των Πρασίνων και EFA. Κυρία υποψήφια Επίτροπε, είπατε ότι χρειάζεστε φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες. Όπως πάμε όμως θα είναι λιγότερες οι επενδύσεις μέχρι το 2030 στις ανανεώσιμες ενέργειες από ότι μεταξύ 2010 και μέχρι 2020. Θεωρείτε ότι πρέπει να μειώσουμε τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες ισχυριζόμενοι ταυτόχρονα ότι θα γίνουμε και το νούμερο ένα στον κόσμο. Δεύτερη ερώτηση. Η Ενεργειακή Ένωση πάνω πει και σύγκληση. Ελπίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό. Ότι χρειάζεται σύγκληση των χωρών. Έχουμε μια οδηγία για τις ανανεώσιμες ενέργειες που είναι και μοχλός για την σύγκληση. Γιατί κάθε χώρα μέλος έχει δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Θα χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα πρωτοβουλίας που θα διαθέτετε ως επίτροπος για να βάλετε δεσμευτικούς, εθνικά δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες ενέργειες και μια σύγκληση των χωρών. Έληξε ο χρόνος σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, αξιότιμε βουλευτή. Πραγματικά πιστεύω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Πράγματι όμως, η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει μια νυχτή. Πιστεύω ότι ο στόχος που δεν είναι το 27% αλλά τουλάχιστον 27% είναι στόχος που θα στηρίξουν ευχαρίστως τα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι αυτό το μήνα θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα κάνουν τον στόχο αυτό του τουλάχιστον 27% δεσμευτικό. Βεβαίως υπάρχει και ο καθορισμός του ενεργειακού μείγματος. Εκεί τα κράτη-μέλη είναι ανεξάρτητα. Αυτά θα αποφασίσουν ποια πηγή ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί. Είναι νομίζω απαραίτητο να υπογραμμίσουμε το εξής. Δεδομένου ότι δεν μπορούν οι λεγόμενες κακές πηγές ενέργειας να υποκατασταθούν μια ανοιχτή. Αυτές που θα διατηρηθούν, ας πούμε, τα, οι ε, υδρογονάνθρακες, είναι πηγές ενέργειας στις οποίες γίνεται τεχνολογική πρόοδος. Πράγμα που σημαίνει ότι η ρήπανση είναι όσο το δυνατόν λιγότερη κατά τη χρήση τους. Στα κράτη-μέλη όσον αφορά την κατάσταση του ενεργειακού μείγματος και την ε, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι ίδια. Είναι λοιπόν δύσκολο να καθορίσουμε ενιαίους στόχους σε εθνικό επίπεδο για όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Προτινόμενη Επίτροπε. Ο κύριος Ντάριο Ταμπουράνο ε, έχει επόμενη ερώτηση. Χαίρετε κυρία Επίτροπε. Ο, λόγο, όρος ε, ε, ανθεκτικότητα χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά και τη χρησιμοποιήσατε και εσείς ε, στα θέματα ενεργειακής απόβασης. Κατά την άποψή μου αυτό το θέμα της ανθεκτικότητας έχει ε, γίνει μια ανθεκτικότητα από πάνω προς τα κάτω. Ε, εστιαζόμαστε περισσότερο σε περισσότερους αγωγούς, σε περισσότερους ε, αγωγούς φυσικού αερίου, ίσως και περισσότερη πυρηνική ενέργεια. Αλλά δεν βλέπουμε τι έχουμε προς τα κάτω ως προς την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος ε, στις τοπικές κοινωνίες οι οποίες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ε, οδεύουμε προς μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση η οποία θα είναι και κατά πάσα πιθανότητα μόνιμη. Σας ε, το ρωτάω αυτό γιατί μάλλον ο όρος δεν είναι και τόσο γνωστός ε, σε άλλους εκτός ευρωπαϊκών οργάνων. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε λοιπόν στους Ευρωπαίους πολίτες πώς ε, νοείτε εσείς την ανθεκτικότητα και πώς μπορούμε να έχουμε συμμετοχή και προς τα κάτω της τοπικής κοινωνίας και της περιφερειακής κοινωνίας στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πράγματι, έχουμε ένα όραμα ανάπτυξης μιας ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης. Η ενεργειακή μας πολιτική πρέπει να ανθέξει στο μέλλον. Αν θέλουμε να έχουμε μια ανθεκτική πολιτική πρέπει να κινηθούμε σε διαφορετικούς τομείς. Το κυριότερο, όταν μιλάμε για ασφάλεια και ήδη το είπα αυτό προηγουμένως πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η εσωτερική αγορά μας θα είναι ισχυρότερη. Θα πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα από ό,τι λειτουργεί. Δεύτερον, εντός της Ευρώπης, εντός της Ενεργειακής Ένωσης, πρέπει να παράγουμε και εμείς ανεξάρτητα περισσότερη ενέργεια. Αυτό θα μας βοηθήσει να μειωθεί η εξάρτησή μας από τις εισαγωγές. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα και όταν μιλάμε για την παραγωγή ενέργειας, στην ουσία μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχουν στην Ευρώπη. Και υπάρχει και κάτι άλλο που σήμερα δεν ανέφερα. Την ενεργειακή απόδοση. Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης τα περισσότερα μπορεί να επιτευχθούν σε τοπικές κοινωνίες, σε τοπικές κοινότητες. Παραδείγματο χάρη, η ανακαίνιση των κτηρίων μπορεί να έχει πολλαπλές επιπτώσεις δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πράσινες θέσεις εργασίας, μείωση των αερίων θερμοκηπίου, μείωση της χρήση της ενέργεια και άρα μείωση της εξάρτηση μας από τι εξωτερικέ πηγές, από ξένους προμηθευτές. Και όλα αυτά αποτελούν μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση. Αυτό θα είναι η ενεργειακή ένωση. Κυρία, ε, κυρία μου, αυτό, ε, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων ε, από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Περνάμε στο δεύτερο γύρο από την κυρία Φρανσουάς Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου και υπάρχει και η πυρηνική ενέργεια η ε, Γαλλία έχει το σύμφωνο πυρηνικής ενέργειας που έχει, ε, την έχει οδηγήσει στη μείωση της ενεργειακής της εξάρτησης στο 50% και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ε, αναπτύξει την πυρηνική ενέργεια και έχουμε μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτή απαιτεί υψηλού επίπεδου θέσεις εργασίας και τεχνολογία καινοτομία κυρία ε, προτινόμενη επίτροπε, πώς θα προχωρήσετε στην αποστολή σας σεβόμενη τη συνθήκη Ευρατόμ η οποία διαρκώς αμφισβητείται από πολλούς. Εσείς κυρία υποψήφια Επιτροπή, ευχαριστώ για την ερώτησή σας κυρία Ευρωβουλευτά. Ίσως επαναλάβω κάτι που δήλωσα προηγουμένως, αλλά οι χώρες μέλη φέρουν οι ίδιες την ευθύνη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ρύθμιση του ενεργειακού τους μίξ και στην χώρα μου, τη Σλοβενία, διαθέτουμε πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μέγα μέρος του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουμε το λαμβάνουμε από αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο. Όταν κληθούμε να ομιλήσουμε περί πυρηνικής ενέργειας θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να θεσπίζονται προδιαγραφές ασφάλειας τις οποίες διαθέτουμε ήδη. Υπήρξαν και ατυχήματα και μετά από τα ατυχήματα που γνωρίζετε, έγιναν δοκιμασίες αντοχής σε όλους του πυρηνικού σταθμού στην Ευρώπη για να γνωρίζουμε αν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές. Εν ώψη της νομοθεσίας που διαθέτουμε, αυτό μπορεί να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλωστε αυτό πρέπει να κάνει προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ κυρία μου. Θα ακολουθήσει ο κύριος Ζιλ Παρνιού Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία υποψηφία επίτροπε, παρά τις πρόοδους που έγιναν τα τελευταία χρόνια, η ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα ενεργείας δεν έχει κατακτήσει τους σημαντικότερους στόχους της πρόσβαση σε λογικές τιμές, ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εξασφάλιση της προμήθειας ενέργειας για όλους και όλες τις Ευρωπαίες, μοντέλο διανομής κατευθυνόμαστε προς, και να κατευθύνουμε προς μια ε, οικονομία που να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίων του άνθρακος. Συμφωνείτε με τους στόχους αυτούς. Θα προωθήσετε τους στόχους αυτούς. Η Ενεργειακή Ένωση θα είναι σαν αυτή που προτείνει ο Ντόναλτ Τάσκ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κοινή αγορά για το φυσικό αέριο όπως έχει προτείνει ε, και ο Ζακ Τελόρα αλλά και εσείς πρόεδρε Μπούσεκ για να αναπτυχθεί μια οικονομία και μια κοινωνία βιώσιμες. Ορίστε λοιπόν συγκεκριμένες ερωτήσεις, παρακαλώ να ακούσω συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτά για τις ερωτήσεις σας. Συμφωνώ άλλωστε μαζί σας ότι στόχος μας στην δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης θα πρέπει να είναι να επιτύχουμε μια ενέργεια εξασφαλισμένη και σε βιώσιμες τιμές. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος τα βασικά στοιχεία της Ενεργειακής Ένωσης είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Πρώτα, μείωση της κατανάλωσης. Αυτό θα οδηγήσει, θα συμβάλλει και σε μια αύξηση της ανεξαρτησίας μας, της ενεργειακής μας ανεξαρτησίας. Ενίσχυση της ε, ενεργειακής μας ανεξαρτησίας χωρίς να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας που πρέπει να είναι μια οικονομία η οποία θα εκπέμπει χαμηλά ποσά αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να βελτιώνεται διαρκώς η τεχνολογία και καύσης ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούμε ακόμη και αν στόχος μας είναι να μειωθεί η εξάρτησή μας τότε ερχόμαστε πάλι στο θέμα της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών. Επίσης απαραίτητο είναι να βελτιωθεί η υποδομή μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο περιφέρειες όπως η Βαλτική και η Ιβυρική που αντιμετωπίζουν αδυναμίες. Όπως είπα, άλλα έργα έχουν προχωρήσει περισσότερο στο σχεδιασμό, αλλά λιγότερο. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος ώστε ότι υλοποιηθούν τα διάφορα έργα. Ωστόσο, έχουν δίκιο όσοι λένε ότι πρέπει να ενισχύσουμε και τη στάση μας απέναντι στους διεθνούς μας εταίρους. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλεί με μια φωνή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τζούλη Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Μπράτουσεκ. Παρά κάποιες ε, πολύ σοβαρές και πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Μέχρι τώρα δεν μας έχετε δώσει και κάποια σαφή απάντηση, απλώς κάποιες ε, κενές επαναλήψεις ε, γενικόλογων δηλώσεων. Θέλετε να σας θέσω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και θα ήθελα να μου δώσετε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Λέτε στις ε, γραπτές σας απαντήσεις και σας παραθέτω ότι η ευφυής ε, φορολογική πολιτική με βάση την αρχή ορυπαίνων πληρώνει είναι κάτι το οποίο σας βρήκε στη σύμφωνη και έτσι θέλετε να τα προχωρήσετε. Ίσως έτσι θέλετε να βρείτε και χρηματοδότηση για όλες τις άλλες δεσμεύσεις που κάνετε ή που δεν κάνετε μέσω των γενικεύσεων που μας κάνετε. Ε, Πώς σκοπεύετε να ακολουθήσετε αυτή την, ε, ε, την άγουσα δεδομένου ότι η φορολογία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Αν συνειδητοποιήσουμε όλοι ποιοι είναι οι κοινοί μας στόχοι, που πιο συγκεκριμένα σημαίνει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τους στόχους που έχουμε καθορίσει από κοινού τα τρία θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, θα πρέπει όλοι από εκεί και πέρα να εργαστούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Όταν γίνεται συζήτηση για τις τιμές της ενέργειας. Στην Ευρώπη έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για τη χρήση καθαρής ενέργειας, για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Και οι τιμές της ενέργειας που πληρώνουμε είναι και λίγο υψηλότερες ε, λόγω και της διαφορετικής φορολόγησης. Εάν λοιπόν θέλουμε να επιτύχουμε τους κοινού μας στόχους ε, στον τομέα της Ενεργειακής Ένωσης, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε από αυτού. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι τα κράτη-μέλη ε, μπορούν να καθορίσουν ανεξάρτητα τη φορολογική του πολιτική. Αν όμως ε, θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια ενεργειακή ένωση, θεωρώ ότι πρέπει και μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για τη συγκεκριμένη πτυχή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες θα είναι υπέρ υψηλότερες ε, φορολόγησης για όσους ρηπαίνουν το περιβάλλον και αυτοί οι οποίοι ρηπαίνουν λιγότερο θα πρέπει να έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Όπως είπατε κι εσείς όμως, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών επ' αυτού. Και επαναλαμβάνω ότι αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία στους κοινούς μας στόχους δεν θα είναι και τόσο δύσκολο, αυτό. Ευχαριστώ ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μπράτουσε και σας ευχαριστώ και διότι δέχεστε και τη θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη ανάπτυξη. Για μένα η Ενεργειακή Ένωση στην Ευρώπη αντιμετωπίζει τρία βασικά προβλήματα. Είναι πολύ ακριβή, ε, ρηπαίνει πολύ και εξαρτώμαστε πολύ από άλλες πηγές. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη μετάβαση της, στη αλλαγή στην ενέργειά μας. Χρειαζόμαστε περισσότερες ανανόησιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτό θα είναι ηράκλειο έργο. Και αυτό είναι σαφές. Συμφωνείτε με αυτή την ανάλυση. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και δεύτερον, Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε επαρκή υποστήριξη από τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό, διότι η Ενεργειακή Ένωση σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ στενή η συνεργασία και αυτό υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τομέα αυτό. Yeah. Ε, ναι, σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε για το ερώτημά σας. Αν έχουμε και πιστεύω ότι έχουμε τους ίδιους στόχους σε σχέση με την Ενεργειακή Ένωση, δεδομένου ότι τους στόχους μαζί τους θέσαμε, ελπίζω ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί. Είπατε ότι θα είναι δύσκολη η συνένεση και η εξέβρεση λύσεων. Συμφωνώ μαζί σας. Η Ενεργειακή Ένωση είναι ότι δεν είναι όσο πιο καθαρή που υπάρχει και ότι έχει μεγάλη εξωτερική εξάρτηση. Τώρα όραμά μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τρία ζητήματα. Αν θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας, πρέπει να παράξουμε περισσότερη ενέργεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από δικούς μας πόρους, είτε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όσο δυνατόν περισσότερο, Επίσης, στην όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση των ορυκτών καυσίμων με τεχνολογίες που θα μολύνουν το περιβάλλον όσο το δυνατόν λιγότερο, που θα ρηπαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο. Κατόπιν, ενεργειακή απόδοση. Με το να είμαστε αποδοτικοί θα μειώσουμε τη χρήση ενέργειας αλλά και την εξάρτηση από τις εισαγωγές. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι το εξής σε όλα τα έργα που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και ανεξαρτησία, ενισχύουμε την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Αυτό έχει αποδειχθεί και πιστεύω ότι αποτελεί κοινό μας στόχος. Η τιμή που πληρώνουμε για την ενέργεια μπορεί να μειωθεί. Γι' αυτό είμαι πεπισμένη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται καλύτερη υποδομή. Sorry, Η κυρία Μέρια Κελόνεν. Κύριε υποψήφια την Πρόεδρε, για να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους πρέπει να προχωρήσουμε προς μια πολιτική ενεργειακού ηλεκτρικού δικτύου που θα επιτρέπει την παρακολούθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή μέχρι την τελική κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο. Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο ευφυές ενεργειακό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Όπως σας είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία, εγώ θα προσπαθήσω να πετύχω το μεγαλύτερο πακέτο των επενδύσεων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ να κατευθυνθεί στον τομέα της ενέργειας και της παραγωγής ή προμήθειας ενέργειας. Ένα μέρος αυτού θα στραφεί και προς τα λεγόμενα έξυπνα δίκτυα. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε και είμαι βεβαία ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είπατε πρέπει να, έχουμε θεοί δίκτυα, έξυπνα δίκτυα, που θα επιτρέπουν στην ενέργεια που παράγεται σε μια άκρη της Ευρώπης να φτάνει τους καταναλωτές στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Για μένα είναι δύσκολο να απαντήσω επακριβώς στο ερώτημά σας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, πότε περιμένουμε να υλοποιηθούν τα έργα αυτά από ό,τι γνωρίζω. Κάποια από αυτά τα έργα είναι πιο προχωρημένα στην προετοιμασία, αλλά όχι τόσο πολύ. Είμαι όμως βεβαία ότι τα έργα που έχουν ήδη προχωρήσει θα στηριχθούν περισσότερο, ενώ άλλα θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπατε και εσείς, τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την επιθυμία μας να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους ανανεώσιμους πόρους είναι απολύτως απαραίτητα. Και γι' αυτό θα φροντίσω να εξασφαλίσω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του προηγούμενου πακέτου επενδύσεων θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Κύριος Βάς Εκόλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπράτουσεκ. Είμαστε εδώ στην Ακρόαση γιατί θα είστε αντιπρόεδρος της Επιτροπής με ευθύνη την Ενεργειακή Ένωση. Αφού ακούσαμε ότι όλα είναι δύσκολα κλπ. κλπ. Αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά θέλουμε να έχουμε έναν αντιπρόεδρο που θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα είναι ισχυρός. Θα ήθελα να είστε πιο σαφείς για το τι θέλετε εσείς, αντί να μας ε, εξηγείτε τη γενική κατάσταση. Ο κόσμος είναι δύσκολος και θέλουμε κάποιον να προχωρήσει την κατάσταση. Όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, ε, θα είσαστε εσείς αυτή που θα είναι επικεφαλής στο ε, διαπραγματεύσει αυτές και βεβαίως τι θα κάνετε για να πετύχουμε το, το στόχο πάνω από 40% στο 2030 γιατί αυτό είναι μικρό, ε, χαμηλός στόχος. Τι θα ε, κάνετε για να πετύχουμε υψηλότερο επίπεδο, πιο φιλόδοξο στόχο. Ευχαριστώ. Η απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτά. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι από μόνη μου δεν μπορώ να επιτυχώ στόχους. Γι' αυτό και τονίζω ότι είναι απαραίτητο οι χώρες μέλη να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων. Πάντως εγώ θα αναλάβω πρωτοβουλίες και θα πράξω τα αναγκαία ώστε να θεσπιστούν φιλόδοξοι στόχοι, αλλά από την άλλη μεριά και ρεαλιστικοί. Θεωρώ σημαντικό να φροντίσουμε να συνεργαστούν, να συμπορευτούν μαζί μας και οι εταίροι μας και εννοώ ιδίως τις Ενωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Γιατί η Ευρώπη όσο φιλόδοξους στόχους και να βάλει, μόνη της δεν μπορεί να αναλάβει, να επομιστεί όλη την προσπάθεια. Ούτε μπορεί να διασώσει το κλίμα μόνη της εφόσον άλλοι εξακολουθούν να ρηπαίνουν με τους ίδιους ρυθμούς. Θα αναλάβω πρωτοβουλίες, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Γνωρίζω πού βρίσκονται και τα όρια, βέβαια και η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν έχει περιορισμούς. Σημαντική είναι η συνεργασία, η συνεργασία με τις χώρες μέλη. Γι' αυτό είπα ότι ελπίζω ότι θα αντιληφθούν οι χώρες μέλη ότι πρόκειται για κοινού στόχους και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνη της δεν μπορεί να τα επιτύχει αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πεντιτσίνη της ομάδας EFDD. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Αντιπρόεδρε, σε όλες τις ακροάσεις, ακόμα και εδώ σήμερα, κάθε φορά που μιλάμε για την ενέργεια, πιο συχνά χρησιμοποιείται ο όρος ενεργειακό μείγμα και βιωσιμότητα. Αυτοί οι όροι δεν είναι πάντα συμβατοί μεταξύ του και ειλικρινά εγώ θεωρώ ότι πίσω από το ε, θέμα του ενεργειακού μείγματο υφέρπει η δυνατότητα που δίνουμε στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν μη βιώσιμε ενεργειακέ πηγέ, όπω γίνεται για παράδειγμα με τα ορυκτά καύσιμα. Να σας πω ότι οι κράτη-μέλη έχουν ήδη εγκρίνει νόμους και διατάξεις που επιτρέπουν ε, μεγαλύτερη χρήση ορυκτών και ε, καυσίμων και μειώνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι μελη δεν ενδιαφέρονται καθόλου αν υπάρχουν ε, απαράδεκτες εκπομπές, γιατί ούτως ή άλλως ε, ε, φορολογούν περισσότερο τους πολίτες για να πληρώσουν το τίμημα. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν σε περίπτωση που υπάρχουν παραβιάσεις από πλευράς κρατών μελών για να υπάρχουν κυρώσεις και να μην είναι πάντα ένοχοι οι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντησή σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αναγκάζομαι να επαναλάβω τα ίδια βέβαια, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι μας ενώνει μια συνθήκη. Και όντως τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε ούτε να αγνοήσουμε, αλλά ταυτόχρονα κάθε κράτος μέλος πρέπει να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να συνεισφέρει στους κοινούς στόχους που έχουμε προκαθορίσει. Σε αυτές τις δύο εβδομάδες προετοιμασίας μου διαπίστωσα ότι όσον αφορά τους στόχους 20-20-20 ε, είμαστε στο σωστό δρόμο. Και όπως είπαν ε, και οι εμπειρογνώμονες, οι στόχοι θα υλοποιηθούν. Δεύτερον, δεν μπορεί να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό και για τις χώρες που ακόμα χρησιμοποιούν ε, ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση της τεχνολογίας ώστε η χρήση των ορυκτών καυσίμων να μολύνει, να ρηπαίνει το περιβάλλον όσο το δυνατόν λιγότερο. Αυτή πρέπει να είναι οι δύο στόχοι μας και να πρέπει να είναι κοινή. Ευχαριστώ πολύ κυρία υποψήφια Αντιπρόεδρε, ο κύριος Σαφχάουζερ έχει το λόγο. Ναι, καλημέρα σας. Πρώτη ερώτηση. Στην ενεργειακή πολιτική, χωρίς τα κράτη έθνη, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πώς προβλέπετε λοιπόν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών εθνών, κυρίως ε, στα μεγάλα έργα για την ε, οικονομία της ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεύτερον, αναφερθήκατε σε 400 δισεκατομμύρια ε, εισαγωγών. Ε, αυτά τα στοιχεία έχω και εγώ. Αν θέλουμε να κάνουμε 10% εξοικονόμηση ενέργειας σε επενδύσεις οι οποίες είναι αποδοτικές σε ε, ορίζοντα 10 ετών θα πρέπει να επενδύσουμε 400 δισεκατομμύρια. Πού θα τα βρείτε εσεί αυτά τα 400 δισεκατομμύρια που αρκετοί αναφέρονται σε 300 δισεκατομμύρια του κ. Γιούνκερ αλλά πολλαπλασιάζονται κάθε φορά που ακούμε κάποιον επίτροπο να μιλάει. Εσεί λοιπόν τα έχετε δει, πού είναι αυτά τα χρήματα. Τρίτον, Έχουμε προτείνει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία ε, από τα, ε, με την υποστήριξη των, ε, του Ταμείου Παρακαταστικών της Γαλλίας και της Ιταλίας προτείνουν κάποια μέτρα επενδύσεων. θα τα υποστηρίξει αυτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Την απάντησή σας παρακαλώ κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όχι, δεν είναι αλήθεια ότι είπα ότι ως αντιπρόεδρος δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα. Πάντοτε όμως υπογραμμίζω και επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της, χωρίς τη συμμετοχή των κρατών μελών, δεν θα μπορέσει να πετύχει και ελπίζω. Δεν ελπίζω, πιστεύω και είμαι σίγουρη, είμαι βεβαία ότι τα κράτη-μέλη το γνωρίζουν αυτό, συγκεκριμένα. Όταν θέτουμε στόχους αποδεχόμαστε και κάποιες δεσμεύσεις. Αυτό είναι όλο. Καθόλου δεν είπα ότι ως αντιπρόεδρος δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Όχι, αλλά αυτό το οποίο σαφώς χρειαζόμαστε είναι η κατανόηση, η συνεργασία και η συμμετοχή των κρατών μελών. Όσον αφορά τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, Εάν θέλουμε μια ισχυρότερη εσωτερική αγορά, ένα στόχος που νομίζω είναι κοινό για όλους μας, αν θέλουμε η ενέργεια να είναι φθηνότερη, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας, τότε πράγματι χρειαζόμαστε σοβαρά ποσά για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Ένα μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα πρέπει να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, ιδιώτες επενδυτές. Αλλά είμαι πεπισμένη, δεδομένου ότι όλοι μας είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, επειδή όλοι μας πιστεύουμε ότι αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη την επόμενη πενταετία, είμαι βεβαία ότι ως εκ τούτου εμείς στο εσωτερικό της Κομισιόν θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις στην Ενεργειακή Ένωση αποτελούν επενδύσεις στις πράσινες θέσεις εργασίας και την πράσινη ανάπτυξη. Αλλά φυσικά η συμφωνία αυτή πρέπει να επέλθει μέσα στην Κομισιόν και συμφωνώ μαζί σας για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και διακόπτει ο Πρόεδρος. Επόμενη ερώτηση, κυρία Έστερ Ντελάνγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ελπίζω ότι την ερώτηση θα την κάνω με το ε, απαλό άγγεγμα της γυναίκας. Φυσικά κυρία Μπράτουσεκ σας συγχαίρω για την υποψηφιότητά σας ως Επιτρόπου για την Ενεργειακή Ένωση και Ενδεχομένως είναι λίγο ηρωνία που εσείς που λέτε ότι σώσατε την, Ευρωπαϊ... Σλοβενία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είσαστε υπεύθυνοι για ένα χώρο που χρειάζεται όπως λέτε περισσότερη Ευρώπη. Όμως ας μην ε, ε, κρίνουμε χωρίς να σας ακούσουμε. τι πρέπει να γίνει και από τα 28 κράτη-μέλη στον τομέα της Ενεργειακής Ένωσης και τι θα μείνει στο κάθε κράτος μέλος τους τρεις πυλώνες. Ποια είναι η πρωτοβουλία που ανυπομονείτε να προωθήσετε, ποια είναι η πιο προσφυλή σας, τι μπορούμε να περιμένουμε, τι είδους αντιπρόεδρες πραγματικά θα είστε. Γιατί νομίζω ότι μιλώ εκ μέρους των περισσότερων εδώ. Πρόσφατα δεν ε, μπορούμε να, δούμε, να ακούσουμε τίποτα παραπάνω από τις τυπικές απαντήσεις. Η απάντηση. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμη κυρία Ευρωβουλευτή, θα, σας πω το εξής. Δεν έσωσα τη Σλοβενία από την Ευρώπη. Έσωσα την Ευρώπη από ένα ακόμα πρόβλημα. Τα περίφημα ντόμινο των αγορών ή αν θέλετε τα χρηματοοικονομικά προβλήματα των κρατών μελών σταμάτησαν στη Σλοβενία. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχει η Ευρώπη ένα μηχανισμό που να βοηθά τα κράτη-μέλη ε, με αλληλεγγύη μεταξύ τους, αλλά είμαι πεπισμένη ότι είναι πολύ καλύτερο και για την ίδια την Ευρώπη, εάν τα κράτη-μέλη είναι σε θέση και μπορούν να λύσουν από μόνο τους τα προβλήματά τους. Ένα, ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι όχι μπορούμε μόνο να συμφωνήσουμε, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε, το οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε στην Ενεργειακή Ένωση, είναι το θέμα της ασφάλειας και το θέμα της, του πώς θα αντιδράσουμε στα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ένα από τα πρώτα μου καθήκοντα, όπως είπα, θα είναι να προετοιμάσω ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης που θα καθορίζει τι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη όταν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις. Η Ενεργειακή Ένωση δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης, αυτό το οποίο συνήθως αναφέρεται. Κατά την άποψή μου, η Ενεργειακή Ένωση είναι και θέμα ευθύνης. Ευθύνης όταν χρειάζεται βεβαίως. Οπότε η Ενεργειακή Ένωση σαφώς είναι ένας χώρος όπου πρέπει πιστεύω να επέλθει συμφωνία και είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Edward. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Έντουαρτ Μάρτιν. Κύρια Μπράτουσεκ, ωραία, Ενεργειακή Ένωση. Αυτό το τίτλο έχει και το χαρτοφυλάκιό σας. Επιμένω τώρα. Δεν έχει ακόμα ουσία αυτό. Μέσα στην οπτική αυτή. Με ποιο τρόπο, συγκεκριμένα θα συμφιλιώσετε τις εθνικές κυριαρχίες του 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ένωσης και από την άλλη μεριά την απαραίτητη σύγκληση που σημαίνει μια κοινότητα της ενέργειας. Θα θέσετε και σε εφαρμογή την τρίτη δέσμη μέτρων που προβλέπει και άλλους τρόπους εκτός από αυτούς που παγορεύουν οι αγορές. Και ποιους. Και ως αντιπρόεδρος θα αγωνιστείτε κατά της ενεργειακής αβεβαιότητας και θα είστε υπέρ της ενεργειακής θωράκισης έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε ένα ελάχιστο ποσοστό ενέργειας και οι πιο στερημένοι συμπολίτε μας. Ευχαριστώ κύριε Μαρτέν, Ευχαριστώ και Ευρωβουλευτά για τις ερωτήσεις σας. Η δημιουργία της Ενεργειακής Ενώσεως, όπως είπα ήδη απαντώντας σε προηγούμενη ερώτηση, θα βασίζεται σε τρεις τουλάχιστον πυλώνες. Πρώτα, στη δημιουργία ή την εξασφάλιση λειτουργίας μιας ισχυρότερης ενιαίας αγοράς και για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε και επέκταση των υποδομών για να καλυφθούν τα κενά, χρειαζόμαστε διαδικτύωση των χωρών μελών, διαδικτύωση μεταξύ των περιφερειών, χρειαζόμαστε δημιουργία δικτύων και μέσα στην ίδια τη χώρα μέλος, εφόσον δεν υπάρχουν, με την βελτιωμένη λειτουργία της ενιαίας αγοράς είμαι πεπισμένη ότι θα κατορθώσουμε να επιτύχουμε ανταγωνιστικότερες τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη προς όφελος και των πολιτών και της οικονομίας. Εισαγωγικά σημείωσα ότι ως πρωθυπουργός της πατρίδας μου φρόντισαν για την πλήρη εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλες τις χώρες μέλη. Βέβαια θα υπάρξουν εξαίρεσεις, αλλά πιστεύω ότι η τρίτη δέσμη μέτρων ενέργειας οφείλει να εφαρμοστεί από όλες τις χώρες μέλη οι κανόνες που περιλαμβάνει το τρίτο αυτό πακέτο μέτρων θα μας επιτρέψουν να ανοίξουμε τις ενεργειακές μας αγορές. Κάτι που θα οδηγήσει σε ευθυνότερη ενέργεια. Ευχαριστώ. Ο Ashley Φοξ. Καλησπέρα κυρία Μπράτουσεκ. Λίγα φαίνεται να γνωρίζετε περί ενεργειακής, ενεργειακής ένωσης. Να σας ρωτήσω κάτι που πάνω θα το ξέρετε. Είπατε στην εναρκτήρια δήλωσή σας ότι εμφανίζεστε ενώπιόν μας εν ταπεινοφροσύνη. Δεν μου φαίνεται σωστό να χαρακτηρίζεστε έτσι με ένα 4% στην ε, χώρα σας δεχθήκατε τα γίνεται υποψήφια να, γίνετε, να, υπο, να υποβληθεί η υποψηφιότητά σας ως επιτρόπου της Σλοβενίας. Ταυτόχρονα γίνονται έρευνες για σας. Δεν έχετε μάλιστα καν δεχθεί τις προσκλήσεις για την έρευνα. Δεν είναι ορθό για μας να γνωρίζουμε τι λέει η έκθεση της Επιτροπής Διοντολογίας του Κοινοβουλίου σας πριν να αποφασίσουμε αν θα γίνετε επίτροπος ή όχι. The please. Ευχαριστώ. Απαντήστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και πάλι την ευκαιρία να σας πω λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία αυτή που αφορά τον ε, ορισμό των υποψηφίων επιτρόπων στη χώρα μου. Ε, θα συμφωνείτε φαντάζομαι μαζί μου ότι η Σλοβανία δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου προκειμένου να ε, υποβάλει κάποιες υποψηφιότητες. Η νέα μας κυβέρνηση ορκίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου και ε, καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε να μην έχει υποβάλει υποψήφιο γέρος η Σλοβενία στον κύριο Γιούγκερ υποβάλαμε ένα κατάλογο με τρία ονόματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και το δικό μου. Και ο κύριος Γιούγκερ από εκεί και πέρα επέλεξε εμένα ως υποψήφια. Ε, από εκεί και πέρα θα πρέπει να τον ρωτήσετε αυτόν για ποιο λόγο επέλεξε εμένα, αλλά εγώ τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που έδειξε το πρόσωπό μου. Η νέα κυβέρνηση δεν ξεκίνησε κάποια διαδικασία διερεύνησης υπόθεσης. Η Επιτροπή κατά της διαφθοράς στη Σλοβενία αποφάσισε ότι ε, λόγω των δημοσιευμάτων στον τύπο θα ξεκινήσει ε, μια διαδικασία για τον έλεγχο της διαδικασίας ορισμού ε, υποψηφίου επιτρόπου. Εγώ είμαι άνθρωπος που ανέκαθαν σεβόμουν τον νόμο, ποτέ δεν είχα προβλήματα με τον νόμο και το χειρότερο το οποίο έχω κάνει είναι να πάρω κλίση για παράνομη στάθμευση. Και κάποια στιγμή στη ζωή μου πήρα και κλίση για υπερβολική ταχύτητα. Δεν ε, ε, μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα η αναθεώρηση της όλης διαδικασίας, βάση και της ε, κείμενης νομοθεσίας, έλαβα την επιστολή ε, που με απευθύνθηκε και έκανα από εκεί και πέρα ό,τι απαιτεί ο νόμος. Πρέπει να σας πω ότι πόρο απέχει η πραγματικότητα από αυτά τα οποία λέγονται, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία ε, έχει οποιαδήποτε ε, στοιχεία διαφθοράς και είναι όλα ασύστολα ψεύδι. Ευχαριστώ. Κυρία Μπράτουσεκ. Άκουσα με χαρά τις παρατηρήσεις σας για το θέμα της ε, βιώσιμης ανάπτυξης και επίσης με χαρά άκουσα τις παρατηρήσεις σας για τη σημασία των πράσινων θέσεων εργασίας. Αναγνωρίζετε λοιπόν τι δυνατότητες υπάρχουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας, το οποίο, ε, ένας τομέας ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικός. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς είναι πώς εσείς ως Αντιπρόεδρος και ε, Επίτροπος Ενεργειακής Ένωσης θα διασφαλίσετε τη συνέχεια της μακροπρόθεσμης μετάβασης σε ουδετερότητα διοξιδίου του άνθρακα, ε, αυξάνοντας ε, ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια ε, βραχυπρόθεσμα, που είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε περισσότερο αυτή τη στιγμή. Πέστε μας επίσης δύο λόγια παραπάνω για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κατανάλωσης και της προμήθειας μέσω ενίσχυσης της νομοθεσίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Την απάντησή σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Συμφωνώ με αυτούς που ισχυρίζονται ότι οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής συμβαδίζουν με τους στόχους που αναφέρατε εσείς. Και το είπα και αρκετές φορές σήμερα. Κάθε φορά που γίνεται μνήα στην ενεργειακή ασφάλεια, πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνουν ταχύτατα, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να είναι πιο μακροπρόθεσμα. Θα μπορούσαν ίσως να είχαν γίνει αρκετά στο παρελθόν και ίσως θα έπρεπε να είχαν γίνει αρκετά στο παρελθόν. Αλλά μετά από την πιο πρόσφατη κρίση φυσικού αερίου, φαίνεται ότι ξεχάσαμε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και αυτό φυσικά με φαίνει και πάλι στο θέμα των υποδομών, που θα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για μας ε, στο επόμενο διάστημα. Και όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναφέρθηκα ε, νωρίτερα στα λεγόμενα ευφυή που είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να μπορούμε να έχουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκεί που την χρειάζονται οι καταναλωτές. Η ενεργειακή δέσμη μέτρων που μας περιμένει, όπως σας είπα, είναι ένα αρκετά μεγάλο πακέτο και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι, δεδομένου ότι όλοι μας ε, θέλουμε να έχουμε πράσινη ανάπτυξη, ένα πολύ μεγάλο τμήμα αυτής της δέσμης μέτρων, αξίας 400 ε, δισεκατομμυρίων, θα ε, πάει σε επενδύσεις οι οποίες ε, θα οδηγήσουν σε καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής μας αγοράς και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού μας τομέα. Η Κορνίλια Ένστ για την επόμενη ερώτηση. <coughs> Κύριε Μπράτουσεκ, βρίσκω ότι είστε πρωταθλήτρια της γενικολογίας. Καλά θα ήταν κάπου κάπου να δίνετε και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα σας δώσω δύο ευκαιρίες. Πρώτη, στα πλαίσια της οικονομικής και νομισματικής κρίσης, πολλές χώρες μέλη μείωσαν τους προϋπολογισμούς τους και για την ενέργεια, όπως Ελλάδα και άλλες χώρες, για διαφόρους λόγους, μειώθηκαν οι τιμές στήριξης, κάτι το οποίο οδήγησε και σε μείωση της χρήσης των ανανεώσιμων ενεργειών. Ερώτηση λοιπόν, ποιες συγκεκριμένε πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για να αναστρέψετε την πορεία αυτή σε αυτές τις συγκεκριμένες χώρες μέλη. Δεύτερο ερώτημα, επίση σημαντικό. Τι θα κάνετε για να είναι προσιτές οι τιμές της ενέργειας για τα νοικοκυριά. Παρακαλώ απαντήστε. Κοιτάξτε, ίσως να, να επαναλάβω πράγματα που έχω πει. Αλλά η αγορά της ενέργειας πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα και θα λειτουργήσει καλύτερα εάν εφαρμόσουμε τα έργα των υποδομών, ε, αν υλοποιήσουμε έργα υποδομών και αν επεκτείνουμε τις υποδομές. Αυτή θα είναι η βάση για να βελτιωθούν οι ροές της ενέργειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μειώσει και τις τιμές και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ήταν το περιεχόμενο της ερωτήσεώς σας. Τώρα για την πρόθεση των ανανεώσιμων ενεργειών Η στήριξη των ενεργειών αυτών για την ώρα είναι στα χέρια των χωρών μελών. Ό,τι ισχύει για την ασφάλεια προμήθειας της ενέργειας ισχύει και για τον τομέα αυτό. Οι χώρες μέλη είναι εκείνες που στο ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλουν να φτιάξουν το πλαίσιο για την στήριξη των φορέων παραγωγής ανανεώσιμων ενεργειών. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα από τα βήματα και ένας από τους στόχους. για την επόμενη πενταετή περίοδο. Είμαι πεπισμένη ότι οι πηγές ανανεώσιμων ενεργειών είναι σημαντικές. Κύριος Έριξον. Είπατε σήμερα ότι ένα μεγάλο μέρος της ενεργειακής πολιτικής βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών. Πράγματι. Όμως Υπάρχουν και πολιτικά εργαλεία που έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτηση, είστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία αυτά τα οποία έχει η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματος χάρη, το Κοινοβούλιο προτείνει υψηλότερους και δεσμευτικούς ε, στόχους για την, για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Είστε διατεθειμένοι να πείτε ναι στο Έτοιμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υψηλότερου και δεσμευτικούς στόχους του κλίματος ή θα τα αφήσετε να ξεφύγει και πάλι αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Η απάντηση παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Με βάση τις σημερινές μου απαντήσεις, διαπιστώνεται ότι οι στόχοι μας για κλιματική αλλαγή είναι σημαντικοί. Έχουμε, πρέπει να θέσουμε φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της δεν μπορεί να δράσει. Χρειαζόμαστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Εάν θέλουμε να υιοθετήσουμε στόχους, πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Επανειλημμένως είπα σήμερα ότι πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Όμως, να μην παραγνωρίζουμε και την πραγματικότητα και τους περιορισμούς που υφίστανται. Επανειλημμένως είπα σήμερα ότι θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, επειδή σαφώς η συνθήκη προβλέπει ποια είναι τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι τα όρια εντός των οποίων τα κράτη-μέλη δρούν ανεξάρτητα. Εγώ είμαι διατεθειμένη να υποστηρίξω υψηλότερους και δεσμευτικούς στόχους σε σχέση με την κλιματική αλλαγή για τους θεωρώ απαραίτητους. Πρέπει όμως ταυτόχρονα όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Δεν έχει νόημα να θέτουμε υπερβολικά ε, φιλόδοξους στόχους αν δεν μπορούμε να τους επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Ο Ρότζερ Χέλμερ. Καλησπέρα, Καλησπέρα σας κυρία Μπράτσεκ. Θα γνωρίζετε κατά πάσα πιθανότητα ότι ο απερχόμενος ε, Επίτροπος Βιομηχανίας, ο κύριος Ταγιάννη, αναφέρθηκε σε σφαγή στην Ευρώπη στη βιομηχανία λόγω αυξαμένων ε, τιμών ενέργειας. Νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα για την ενέργεια, για τη διασύνδεση, για, την, για τον ανταγωνισμό, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι ο βασικός στόχος αυτών των υπερβολικών τιμών είναι η μεγάλη δέσμευση που έχουμε για δαπανηρές ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίση και αυτή η αιμονή που έχουμε με το σύστημα εμπορία εκπομπών. Ε, είστε ικανοποιημένοι να βλέπετε ενεργοβόρε. Ε, ε, βιομηχανίες να φεύγουν τελείως από την Ευρώπη παίρνοντας μαζί τους και τις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις και γνωρίζετε ότι πολύ συχνά πηγαίνουν σε περιοχές τις οποίες υπάρχουν πολύ κατώτερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Αντί να καταστρέφεται λοιπόν απλώς και μόνο θέσεις στην Ευρώπη, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα αυξάνεται και την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας. Ευχαριστώ ε, συνάδελφε η απάντηση παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμε Ευρωβουλευτά. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αναφέρθηκα συχνά στην ανταγωνιστικότητα σήμερα και θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά το εξής. Εάν εμείς δημιουργήσουμε μια ενισχυμένη εσωτερική αγορά, αν ολοκληρώσουμε τις υποδομές, εάν εξασφαλίσουμε ε, ότι θα υπάρχει απρόσκοπτη ε, βίβαση ενέργειας στην Ευρώπη, τότε θα μπορούμε να έχουμε κατάλληλες τιμές ενέργειας και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Θεωρώ ότι αυτό είναι του σημασίας, το πιστεύω ακράδαντα και θεωρώ ότι υπάρχουν και εμπειρίες σε επίπεδο κρατών μελών. Η άξιση της ανταγωνιστικότητας οδήγησε σε μείευση των τιμών ενέργεια. Η Σλοβενία είναι μία από αυτές τις χώρες. Υπάρχει μία έκθεση από την ε, αρμόδια γενική διεύθυνση και εκεί βλέπετε ε, ότι οι τιμές της ενέργειας στη Σλοβενία μειώθηκαν κατά περίπου 30% όταν εισήρθε ένας νέος παράγων στην αγορά της ενέργειας. Αυτό σίγουρα δεν αποτελεί σύμπτωση. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας ε, στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, σίγουρα πρέπει να κάνουμε επενδύσεις και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με περισσότερες επενδύσεις, με μεγαλύτερη ανάπτυξη ε, θα έχουμε ε, φθηνότερες και καλύτερα διαθέσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, έχουν, τιμές, ε, ε, έχουν μειώσει στις τιμές και θεωρώ ότι αυτό είναι ένας τρόπος να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Πρέπει να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να επιτύχουμε τους στόχους μας αυτούς. Τελευταίος ο μιλητής στον τρίτο γύρο ερωτήσεων, ο κύριος Ζανλίκ Σαφχάιουζερ. Ευχαριστώ. Κυρία μου, η ερώτησή μου αφορά τις προτεραιότητές σας. Πιστεύετε απλώς και μόνο στην τέλεια ανταγωνιστικότητα και στην τέλεια αγορά ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δράση από πλευράς κρατών μελών για να μπορέσει να υπάρξει μετεγκατάσταση της ενεργειακής παραγωγής ε, χάρη σε αυτό το οποίο αποκαλούμε το, ε, τα σύντομα κυκλώματα, να έχουμε ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, ασφάλεια εφοδιασμού επίσης. Και αυτό φυσικά θα μπορούσε να ισχύει και για τα μικρότερα δίκτυα αλλά και για την διασύνδεση των δικτύων ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί για να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα κάποια δίκτυα τα οποία θα στοιχίζουν λιγότερο σε ενεργειακό επίπεδο στον αγροδιατροφικό τομέα και στον ε, τομέα της μεταποίησης. Θα μπορούσατε να μας πείτε ε, την άποψή σας για αυτά τα μικρά ε, σύντομα δίκτυα στον ενεργειακό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. απάντηση παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Αξιότιμε Ευρωβουλευτά, είμαι πεπισμένη ότι όπως εγγυάται και η τρίτη δέσμη μέτρων της ενέργειας, η αγορά ενέργειας πρέπει να την χάνει καλής ρύθμισης, καλής νομοθεσίας. Επιπλέον δε, είμαι απόλυτα πεπισμένη και σας το είπα και προηγουμένως αναφερόμενη στην ε, περίπτωση της Σλοβενίας, ότι υπάρχει ακόμα απόθεμα ώστε να φροντίσουμε η ενέργεια ε, για την Ευρώπη ε, να είναι φθηνότερη. Και Όπω επεσήμανα σήμερα και το επανέλαβα αρκετέ φορέ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι μία ισχυρότερη εσωτερική αγορά θα είναι προς όφελος όλων. Γι' αυτό λοιπόν και καθήκον μας τα επόμενα χρόνια θα είναι η ενίσχυση των υποδομών. Δυστυχώς Κάποια σχέδια στον τομέα αυτό είναι πιο προηγμένα σε σχέση με κάποια άλλα που υπολείπονται ε, και δεν θα είναι εύκολο να αλλάξουν τα πράγματα εν μία νυχτή. Αλλά εάν ε, αντιμετωπίσουμε και πάλι κρίση φυσικού αερίου, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να αποφύγουμε να δημιουργηθεί μια ανοιχτή. αλλα εαν αντιμετωπισουμε και παλι κριση φυσικου αεριου οπως σας ειπα και προηγουμενως θα πρεπει να αποφυγουμε να δημιουργηθει μια κατασταση σαν αυτή του 2009 όταν λησμονήσαμε πόσο σημαντικές ήταν οι κατάλληλες υποδομές. Ε, μια ισχυρή εσωτερική αγορά ε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Ολοκλήρωσα εγώ από πλευρά μου ε, και τώρα δίνουμε το λόγο στον ε, Πρόεδρο, στον κύριο Τζοβάνι Λαβία. ευχαριστώ. Η συνάδελφος Σουίτσα για την ερώτησή της τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπράτουσεκ. Επεριλημμένως αναφερθήκατε στην διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Πιστεύω ότι ο, ο ΤΑΠ, ο αγωγός που θα περνάει από την Αδριατική μεταφέροντας φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν θα είναι πολύ σημαντικός δεδομένου ότι μας ενδιαφέρει ο περιορισμός της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο και δεδομένου ότι ε, έχουμε καλή συνεργασία με τη Ρωσία. Σας έχω δει όμως ε, σε ένα βίντεο να μιλάτε εναντίον της Ευρώπης μήπως θα και να τραγουδάτε κομμουνιστικά τραγούδια. Μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε το μέλλον και να ξεχάσουμε τον κομμουνισμό. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευρωβουλευτή. Σας ευχαριστώ που με την ερώτηση αυτή μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω μία απάντηση και να ξεκινήσω από το εθνικό θέμα. Το βίντεο το οποίο είδατε αφορά την ε, τελετή της ε, τελετής για το μέτωπο της ανεξαρτησίας. Το τραγούδι που τραγούδισα και δεν ήταν το μόνο, δεν ήταν αυτό όπως το περι, περιγράφεται. Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρες οι αξίες της Ευρώπης στο χώρο αυτό και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ. είναι ένα αντιφασιστικό ταξίδι. Εγώ δεν ήμουν ποτέ μέλος οποιοδήποτε κομμουνιστικού κόμματος. Στη Σλοβενία έχω επικριθεί για το αντίθετο. Μου ε, με κατηγορούν ότι είμαι υπερβολικά φιλοευρωπαία, ότι ακολουθώ τις επιταγές των Βρυξελών και ότι δεν αντιστέκομαι σε αυτές. Αυτό μου προσάπτουν. Πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι ο σωστός δρόμος για τη χώρα μου και είμαι πολύ περήφανη που η Σλοβενία είναι ενταγμένη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τώρα όσον αφορά τη διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών. Βεβαίως το έργο που αναφέρατε είναι απαραίτητο. Το έργο αυτό εξορισμού θα μειώσει την εξάρτησή μας από τη Ρωσία και θεωρώ ότι όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα στον τομέα αυτό. Άρα πρέπει να πω ότι είμαι υπέρ του έργου αυτού, του αγωγού ΤΑΠ. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους ε, δρόμους που θα μας οδηγήσουν εκεί που επιθυμούν. Ο συνάδελφος κύριος Γκασπάρα έχει δει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε Μπράτσεφ. σας έχει ανατεθεί ένα σημαντικός ρόλος με στρατηγικό και φιλόδοξο στόχο και εξαιρετικό φυσικά αν καταφέρουμε να τον επιτύχουμε, ε, η Ενεργειακή Ένωση. Γι' αυτό και λοιπόν θα ήθελα να με συγχωρέσετε αν επιμένουμε ε, για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς επιθυμάτε από πολιτική σκοπιά και τι πόρους σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για αυτόν τον τόσο σημαντικό στόχο. Αναφερθήκατε σε ένα σημαντικό ποσοστό, σε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των 300 δισεκατομμυρίων για επενδύσεις που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να κατανοήσω λίγο καλύτερα ποια είναι η ποσόστοση τι κομμάτι θα πάρετε εσείς από την τούρτα, τι σκοπεύετε να ζητήσετε, τι σκοπεύετε να δεσμεύσετε από αυτά τα 300 δισεκατομμύρια επενδύσεις, πώς σκοπεύετε να εκμεταλλευτείτε τα διαφορετικά ταμεία, ε, να, να χρησιμοποιήσετε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, προηγουμένως ε, διακόψετε και μας είπατε ότι θα απαντήσετε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ, ο λόγος στην, στην υποψήφια Επίτροπο. Eh, Ευχαριστώ για την ερώτηση. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, που αν δεν απατώμε είναι 284 αυτή τη στιγμή, έχουν συνολική αξία 40 έως 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα μεγάλο ποσοστό θα προέλθει από την οικονομία και από επενδυτές. Το υπόλοιπο είναι επίσης σημαντικό και ένα μεγάλο κομμάτι των 300 δισεκατομμυρίων ελπίζουμε ότι θα κατευθυνθεί στα έργα αυτά. Εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια γι' αυτό. Θα, μου είναι δύσκολο να αναφέρω συγκεκριμένο αριθμό σήμερα, αλλά είμαι πεπισμένη ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι κοινό μας στόχος. Οι νέες θέσεις εργασίας αποτελούν κοινό στόχο και τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έργα τον ενεργειακό χώρο, τα μεγάλα έργα υποδομής, αλλά και άλλα έργα που αφορούν την ε, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, δίνουν θέσεις εργασίας και συνεισφέρουν στην πράσινη ανάπτυξη. Ένα, μια άλλη πηγή, ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και που αφορά την ενέργεια είναι κάτι το οποίο σαφώς θα, θα προσπαθήσω να επιτύχω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόρμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει και το αέριο συστολήθου. Εκεί βέβαια χρειάζεται να υπάρχουν αυστηροί περιβαλλοντικοί έλεγχοι. η εξόριξη του αερίου του σχιστολίθου προκαλεί και ορισμένα, ορισμένες ανησυχίες βέβαια περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Φαίνεται πως το πρώτο από το αέριο αυτό θα αρχίσει να εξορίστε στην Ιρλανδία το 2018 και θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Τι λέτε εσείς τώρα για τις νέες αυτές μορφές ενέργειας, το σχιστολιθικό αέριο καθώς και την ενέργεια των κυμάτων. Ευχαριστώ και Ευρωβουλευτά για τις ερωτήσεις σας. Το σχιστολιθικό αέριο ασφαλώς αποτελεί επιλογή. Μία από τις επιλογές που διαθέτουμε. Εγώ τουλάχιστον είμαι πεπισμένη ότι εφόσον τεθεί το ερώτημα εάν θα χρησιμοποιήσει μια χώρα ή όχι το αέριο αυτό, αυτοι τις αποφάσεις θα πρέπει να προηγηθούν σε βάθος αναλύσεις και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι να διασφαλίσει ότι τηρούνται όλες οι ισχύουσες εκείνη τη στιγμή περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε αυτομάτως να μεταφέρουμε ό,τι γίνεται στις ΗΠΑ και να το εφαρμόσουμε και στην Ευρώπη. Εδώ σε εμά η πυκνότητα πληθυσμού είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό είναι ήδη ένα επιχείρημα που οφείλει να ληφθεί υπόψη για την εκμετάλλευση του αέριου αυτού. Τι επιπτώσεις θα έχει στους υδροφόρους ορίζοντες. Αναλύσεις που πρέπει πρώτα να γίνουν πριν να λάβει την απόφαση μια χώρα μέλος εάν θα χρησιμοποιήσει την επιλογή αυτή ή όχι, του σχιστολιτικό αέριου. Επαναλαμβάνω ότι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άρα και δικό μου θα είναι να διασφαλίσουμε ότι στην περίπτωση ενδεχόμενης χρήσης αυτής της επιλογής η συγκεκριμένη χώρα μέλος τηρεί όλες τις περιβαλλοντικές διατάξεις που ισχύουν. Ο κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε. ως Αντιπρόεδρος ε, υπεύθυνη για την Ενεργειακή Ένωση, πώς θα διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει κατάλληλο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, βάσει και της αποστολής σας. Τι ρόλο βλέπετε να διαδραματίζουν ε, τα προηγμένα καύσιμα στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα. Προς το παρόν η Επιτροπή φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να μας δώσει στοιχεία, αλλά η βιομηχανία θα τα χρειαστεί. Ε, ελπίζω λοιπόν να υπάρχει ένα όσο το δυνατόν σαφέστερο μήνυμα για το μέλλον. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα αρκετέ φορές σήμερα, είναι γεγονός ότι εμείς στην Ευρώπη εξακολουθούμε να εξαρτώμαστε πάρα πολύ από την εισαγωγή ενέργειας. Εισάγουμε περίπου ενέργεια αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα. Αν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε την εξάρτησή μας, ε, που είναι μια εξάρτηση της τάξης του ενός πέμπτου ετησίως, ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε δικούς μας ενεργειακούς πόρους και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σαφώς ε, βρίσκονται σε πληθώρα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν στη λύση. Αλλά και πάλι, και εδώ πανέρχομαι στο θέμα των υποδομών, χρειαζόμαστε υποδομές ώστε η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές να φτάνει μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η δημιουργία των ευφυών δικτύων είναι αυτό το οποίο μας περιμένει στην Ευρώπη, στην Ενεργειακή Ένωση στην επόμενη πενταετία, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε με αποτελεσματικό τρόπο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και πάλι όπως σας ανέφερα σήμερα, οι στόχοι της Ευρώπης 2020 θα επιτευχθούν και όσον αφορά το 2030 Είμαι βέβαιη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία το... εντός του Οκτωβρίου. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, θα φτάσει στο 27% εξ όσων γνωρίζω. Αλλά και πάλι, όπως σας είπα επανειλημμένο σήμερα, το ενεργειακό μείγμα εν τέλει είναι στα χέρια των κρατών μελών. Και Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μόνο από κοινού θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Ο ρόλος ε, στον ε, κύριο Βάουντς. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τον πυρηνικό σταθμό της ε, νουκλεόνιο που βρίσκεται πολύ κοντά στο Μπιλμπάο ε, και στο Μπόργος. Ε, πρόκειται για δύο εργοστάσια, έχουμε δύο εργοστάσια που ήταν της ίδιας τεχνολογίας που έκλεισαν στο Βέλγιο λόγω παροχημένης τεχνολογίας, αλλά το συγκεκριμένο σταθμό είναι ακόμα ανοιχτό και η Ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει τη διατήρηση του, ε, του σταθμού αυτού. ενώ στην αυτόνομη χώρα των Βάσκων είναι κατά η κυβέρνηση. Ε, θα ζητήσετε τουλάχιστον να κλείσουν οι πυρηνικοί σταθμοί που είναι πιο παλιοί και πιο επικίνδυνοι. Δεύτερη ερώτηση όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Επειδή η οδηγία αναγνωρίζει και ε, προτιμά την ε, επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων αντί άλλων τεχνικών παρά το γεγονός ότι είναι πιο δαπανηρή, τι συγκεκριμένες προτάσεις θα παρουσιάσετε ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των αποβλήτων που ανακυκλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το συγκεκριμένο πυρηνικό σταθμό που αναφέρατε, δύσκολα θα σας απαντήσω συγκεκριμένα γιατί δεν γνωρίζω την περίπτωση όμως, θα το μελετήσω και είμαι βεβαία ότι θα μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα συγκεκριμένα κάποια στιγμή. Τώρα, όπως είπαμε προηγουμένως, το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να φροντίσει η πυρηνική μας σταθμή, ενώ η, σταθμή, η πυρηνική σταθμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παραμείνουν ασφαλείς. Εξ όσων γνωρίζω, τα τεστ αντοχής που έγιναν απέδειξαν ότι η πυρηνική μας σταθμή πράγματι είναι ασφαλής. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη έχουμε και μια σειρά από παλαιότερους πυρηνικούς σταθμούς και άρα γίνεται ακόμα πιο σημαντικό να παρακολουθείτε το θέμα της ασφαλείας τους. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, όπως είπατε και εσείς. Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των αποβλήτων και να φροντίσουμε τα επικίνδυνα αυτά απόβλητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά χωρίς να έχουν βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα αυτό, αλλά το κρίσιμο ζήτημα που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο εγώ μπορώ να προσφέρω είναι το θέμα της ασφάλειας και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας τα στοιχεία μέχρι στιγμή έχουν δείξει ότι τα η πυρηνική σταθμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ασφαλής και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Γιάννη Κλιαντόπτου. Ευχαριστώ πολύ. Θα αναφερθώ στο θέμα του κινέζικου dumping στα φωτοβολταϊκά πάνελ. Έχει φανεί ότι αυτά είναι το 50% της ευρωπαϊκής αγοράς και η δική σας κυβέρνηση μαζί με άλλες κυβερνήσεις έδωσαν μάχη για να περιοριστούν όσο δυνατόν περισσότερο τα μέτρα anti-dumping της Ευρώπης απέναντι σε ένα dumping που κατέστρεψε τη σχετική ευρωπαϊκή βιομηχανία, πράγμα που οδήγησε να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Λέτε ότι θα υποστηρίξετε την ευρωπαϊκή βιομηχανία, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά θα υπερασπιστείτε τον τομέα της φωτοβολταϊκής ενέργειας ή θα κάνετε αυτό που κάνουν όλο και περισσότερο σήμερα στην Ευρώπη υπό την ε, επιρροή χωρών όπως η Σλοβενία ε, θα, κάνουν, θα κινηθούν προς την κατεύθυνση που θα, ευχαριστεί, θα είναι ευχάριστη στη σχέση μας με την Κίνα. Ε, Σα ευχαριστώ. για την ερώτηση. Είναι ένα ερώτημα που και εγώ το αντιμετώπισα την εποχή που ήμουν πρωθυπουργός. Τότε που επιδοτήσαμε τη ηλιακή ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι νομίζω σημαντικό να δώσουμε αγώνα για την οικονομία μας, να την υποστηρίξουμε. Όλα όμως αυτά πρέπει να συνάδουν με τους, κανόνες των, τους διεθνείς κανόνες των αγορών. Άρα Δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πεντιτσίνη τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφια Αντιπρόεδρε, κάποιος ε, συνάδελφος ε, πριν από μένα σας έκανε μία ερώτηση για την πυρηνική ενέργεια και εσείς και πάλι απαντήσετε ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν το ενεργειακό τους μείγμα. Εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Να με. Συνεχίζω λοιπόν. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας μιλήσω και πάλι για ε, τα ενεργειακά, τα πυρηνικά απόβλητα. Σας παρακαλώ μην μου λέτε ότι θα λάβετε κάθε δυνατό μέτρο για να έχετε ασφάλεια στην αποθήκευση των ε, αποβλήτων δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζείτε εσείς, αλλά στο δικό μου τον κόσμο υπάρχει μεγάλη διαφθορά και είμαι βέβαιος ότι τα απόβλητα αυτά κατά πάσα πιθανότητα θα θαυτούν κάτω από κάποιον ε, ε, πολίτη και δεν θα τα ανανεω, ε, ανακυκλώσουμε. Πέραν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, τις οποίες μας αναφέρετε συνεχώς, τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για να μην μην υπάρχει πυρηνική ενέργεια μεταξύ των επιλογών του ενεργειακού μείγματος. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όσο την ευθύνη φέρουν οι χώρες μέλη για το ενεργειακό τους μείγμα, και αυτές είναι σύμφωνα με τη συνθήκη οι αρμόδιες. Και για να παρέμβουμε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει τροποποίηση της συνθήκης. Το ίδιο ισχύει άλλωστε και για την πυρηνική ενέργεια. Που και αυτή είναι αρμοδιότητα των χώρων μελών. Σύμφωνα με τη συνθήκη. Καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξάλλου είναι να ερευνά και να εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία των πυρηνικών σταθμών. Είπα και πριν ότι σύμφωνα με τα όσα είπαν οι εμπειρογνώμονες μετά τις δοκιμασίες αντοχής, τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη έχουν καλώ. Ε, δεν πήγα και η ίδια να τα δω. Πιστεύω τους εμπειρογνώμονες που είπαν στις εκθέσεις τους ότι είναι εντάξει. Αυτό είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εξετάζει την ασφαλή λειτουργία τους. Διότι, επιμένω, είναι γεγονός ότι οι ίδιες χώρες μέλη είναι αρμόδιες και αυτές αποφασίζουν σχετικά με το ενεργειακό τους μείγμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Κυρία Υποψηφία Επίτροπε, είπατε κατ' επανάληψη ότι μεγάλη προτεραιότητα θα έχει διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών της ενέργειας. Θέλω να καταλάβω λίγο περισσότερο, διότι ως Πρωθυπουργό νομίζω κάνατε το αντίθετο. Υποστηρίξατε τον αγωγό South Stream κατά του Ναμπούκο που ήταν ευρωπαϊκό έργο και έτσι συμβάλατε στην αύξηση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο εννοείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν γίνετε τελικά επίτροπος, ποια στάση θα τηρήσετε απέναντι στον South Stream και ποια θα είναι η στάση σας απέναντι στον αγώνα Μπούκο. Θα χαρώ πολύ να μου δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση και όχι τύπου προπαγάνδα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω σαφώς. Ο Ναμπούκο ήταν θετικό έργο για την Ευρώπη, καλό έργο, για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας από έναν και μοναδικό προμηθευτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο δεν έκανε τίποτε. Οι επενδυτές θεώρησαν ότι το έργο δεν ήταν ενδιαφέρον για αυτούς και φαίνεται ότι δεν πάει να υλοποιηθεί, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επενδυτές έτσι αποφάσισαν. Σε ό,τι αφορά τον αγωγό South Stream, όντως παίρνουμε το αέριο από τον μοναδικό προμηθευτή από τον οποίο εξαρτώμεθα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι πρέπει να προωθηθεί η διαφοροποίηση και των ροών και ω Πρωθυπουργό της χώρας μου μάλιστα τάχθηκα υπέρ αυτή τη ιδέας και να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες για όλα τα έργα και για τον South Stream όπου και εκεί πρέπει να τηρούνται όλοι οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Αυτό υπεστήριξα και ως Πρωθυπουργό της χώρας μου και αυτό θα υποστηρίξω και ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό και άλλωστε τίποτε άλλο δεν έκανα και ως Πρωθυπουργός. Κάρλος Ζωρίνιο. Πρέπει να έχουμε προφορίες ρεαλιστικές. Η Ευρώπη πρέπει να παίξει ρόλο πρωτοπόρου στις ευφυείς ενέργειες και στα ευφυεί συστήματα ενέργειας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένα όραμα. Και αυτή πρέπει να είναι η βασική αφετηρία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης. Ποια στάση θα τηρήσετε και απέναντι στις διεθνείς αγορές, όπως αγορές τηλεπικοινωνιών, για παράδειγμα. Θεωρείτε ότι μπορεί να κινδυνεύσει η ευρωπαϊκή αγορά. Πώς θα πλαισιώσετε την διαδικασία ώστε μεταξύ άλλων η προσωπική σφαίρα, τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών να μην κινδυνεύσουν. Ja, ε, ε, najlepša hvala tudi za Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την ερώτησή σας. Σήμερα αναφερθήκα αρκετές φορές στο θέμα των υποδομών και την ανάγκη να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επαναλαμβάνω και πάλι, εάν θέλουμε να υλοποιήσουμε το βασικό μας όραμα, δηλαδή μία ενεργειακή ένωση ανθεκτική με πολύ σαφείς ε, στόχους σε θέματα κλιματικής αλλαγής, καθήκον μας είναι καταρχάς η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς το συντομότερο δυνατόν και ταυτόχρονα ε, κάποιος ε, αναφέρθηκε νωρίτερα στο hardware ε, ενώντας τις υποδομές. Συμφωνώ μαζί σας. Χρειαζόμαστε hardware αλλά χρειαζόμαστε και λογισμικό. Χρειαζόμαστε δηλαδή σαφέστερους κανόνες για να διασφαλίσουμε την αγαστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτές οι δύο πτυχές λοιπόν, το hardware και το software, είναι αυτό το οποίο μας αναλογεί για να έχουμε μια ιστορική αγορά που θα λειτουργεί και θα μπορούμε να ε, υλοποιήσουμε τους βασικούς μας στόχους ε, στην Ενεργειακή Ένωση. Μικρότερη εξάρτηση, καθαρότερη ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές. Ευχαριστώ και τώρα ο λόγος του συνάδελφο το Ζενόσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε στις απαντήσεις σας ακούμε συνεχώς ε, ότι η προτεραιότητά σας είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θέλετε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, στο ενεργειακό μείγμα. Αλλά για πολλά κράτη-μέλη η πυρηνική ενέργεια και η ενέργεια από ρηκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ σημαντικές πηγές, ιδίως ο άνθρακας. Υπάρχει λοιπόν ένα παράδοξο εδώ. εκδηλώνουμε με το ενδιαφέρον μας, αλλά η οικονομία μας οδηγεί σε εντελώ διαφορετική συμπεριφορά. Η οικονομία της σήμερων ημέρα δεν μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε κατάλληλες πηγές, ε, βιώσιμες πηγές σύντομα. Είναι ρεαλιστικό λοιπόν αυτό το οποίο μας λέτε ή ε, θα έπρεπε να προσπαθήσετε να είστε λίγο, να είστε λίγο πιο ρεαλίστρια για την ε, εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος. Ευχαριστώ. Σήμερα επανειλημμένος επεσήμενα ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστές. Διότι εάν καθορίσουμε πάρα πολύ φιλόδοξους στόχους τους οποίους στη συνέχεια δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ε, όλο αυτό δεν θα χρησιμεύσει σε τίποτα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα εν μία νυχτή γνωρίζω ότι η κατάσταση πόρα απέχει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Κάποιοι χρησιμοποιούν περισσότερο ρηκτό καύσιμα από άλλους. Ε, κάποιοι έχουν ήδη πολύ υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στο ενεργειακό τους μείγμα. Και θεωρώ ότι ο στόχος και νομίζω ότι επ' αυτού θα συμφωνώ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, είναι να έχουμε τουλάχιστον 27% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Πρόκειται για ένα στόχο, ο οποίος κατά την άποψή μου ε, μπορεί να υλοποιηθεί και ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτυχθούν και νέες τεχνολογίες για τη χρήση των ε, ορυκτών καυσίμων, ώστε να μην είναι τόσο σημαντικές οι συνέπειές τους για το περιβάλλον. δεν θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε από τη μια στιγμή στην άλλη πηγές ενέργειας που είναι πιο ρηπογόνες ε, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα στον τομέα αυτό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα, χρησιμοποιηθούν, θα χρησιμοποιούνται τα ορυκτά καύσιμα με τον πιο καθαρό τρόπο, με τις κατάλληλες τεχνολογίες. Όσον αφορά τώρα την πυρηνική ενέργεια, νομίζω ότι ήδη απάντησα και σας είπα την άποψή μου στις προηγούμενες απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δράσει κυρίως στον τομέα της ασφάλειας. Ευχαριστώ η κυρία Μιλίνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη υποψήφια. Στην επιστολή ανάθεσης ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι θα πρέπει να συντονίσετε διάφορους επιτρόπους μεταφορά ενέργεια, διάστημα και μεταφορές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θαλάσσια ε, πολιτική, ε, αγροτική ανάπτυξη και βεβαίως μεταξύ όλων των άλλων έρευνα και ανάπτυξη. Όλοι μας φοβούμαστε ότι το έργο αυτό είναι τεράστιο. Οπότε σας ρωτώ πώς σκοπεύετε να εξασφαλίσετε ότι ο συντονισμός αυτός θα αποβεί επιτυχημένος. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, κυρία Μλινάρ. Πράγματι, πράγματι, μιλάμε για μια μεγάλη πρόκληση που δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά όλους μας, ολόκληρη την ε, Επιτροπή. Η νέα δομή της Επιτροπής έχει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση και πρέπει να φροντίσουμε ότι η νέα αυτή οργανωτική δομή θα είναι λειτουργική. Όπως είπα και στην εναρκτήρια ομιλία μου, εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος μου είναι να εξασφαλίσω ότι οι διάφοροι στόχοι από διάφορους τομείς θα ενταχθούν σε μια ενιαία στρατηγική με κοινούς στόχους, έτσι ώστε να μην καταλήξουμε να έχουμε αντιφατικούς στόχους σε διάφορους τομείς. Ελπίζω λοιπόν ότι η εμπειρία μου ως Πρωθυπουργού όπου ήμουν επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνασπισμού τεσσάρων κομμάτων, θα μου έχει δώσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να βρω λύσεις που όλοι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Βεβαίως, πολλοί λένε ότι κάποιες θέσεις είναι αδύνατο να συμβιβαστούν. Θεωρώ όμως ότι η εμπειρία μου στον τομέα αυτό θα με βοηθήσει στο έργο του Επιτρόπου αν φυσικά το αναλάβω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκριμπ. Ευχαριστώ κυρία Υποψηφία Επίτροπε. Εδώ με βλέπετε. Είπατε ότι η τρίτη δέσμη μέτρων ενέργειας σας βρίσκει ενθουσιοδός σύμφωνη. Μιλήσατε πολύ και για υποδομές στην ενιαία αγορά. Θεωρείτε ότι αυτό το τρίτο πακέτο ενέργειας, αυτό το πακέτο ενέργειας επαρκεί για να στηρίξει τις επενδύσεις αυτές. Δίκτυα ενέργειας, αγωγούς και πολλά έργα τα οποία ε, δεν έχουν γίνει ακόμη. Δεύτερο, θεωρείτε ότι μπορούμε να βρούμε και άλλες λύσεις πέραν των όσων περιλαμβάνονται στο πακέτο, εννοώ ιδιαίτερα τον ΟΟ South Stream. Και τέλος, σύντομη ερώτηση. Ποια είναι η θέση σας απέναντι στην απαγόρευση επανεξαγωγής του φυσικού αερίου. Πρόσφατα είδαμε αυτές τις απαγορεύσεις επανεξαγωγών που έχουν επιβάλει οι Ρώσοι εταίροι. Ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις σας. Είμαι πεπισμένη ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί πλήρως το πακέτο μέτρων για την ενέργεια. Σε όλες τις χώρες μέλη, χωρίς καμιά εξαίρεση. για όλες τις επενδύσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και ο South Stream θα πρέπει να ισχύουν χωρίς εξαίρεση οι ίδιοι κανόνες. Εξήγησα ότι χρειαζόμαστε και το hardware, δηλαδή τις ε, ε, επενδύσεις και το software, το σχεδιασμό. Για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς χρειαζόμαστε κανόνες που να εξασφαλίζουν τη λειτουργία της αγοράς. Γι' αυτό μίλησα σήμερα πολλές φορές για τις αναγκαίες επενδύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλούμε για μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά. Εγώ δεν είμαι βεβαία ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θέλετε πιο συγκεκριμένα η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να μιλούν με μια φωνή απέναντι σε εταίρους εκτός των συνόρων μας. Άλλωστε θεωρώ σωστό απέναντι στη Ρωσία να μιλούμε με μια φωνή. Και να συμφωνούμε πρώτα μεταξύ μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θέλουμε να προχωρήσουμε και πώς θέλουμε να αντιδράσουμε γιατί αυτός είναι ο μοναδικός ορθός τρόπος αν θέλουμε να είμαστε ισχυρότερος εταίρος απέναντι στους Ρώσους από ό,τι είμαστε σήμερα. Κάθε χώρα μέλος μόνη της είναι πολύ τροτότερη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ενιαία φωνή. Ο κύριος Ντάνς. Καλά λέτε, εδώ είμαι, σηκώνω το χέρι μου να μιλούμε μια φωνή και μιλήσατε και πολύ για ρεαλιστικούς στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει υψηλή προτεραιότητα και στο στόχο προστασίας του κλίματος. Εσείς θα είστε επικεφαλής των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολύ σημαντικές συνομιλίες για την ε, ε, διάσκεψη COP και για τη διάσκεψη των Παρισίων του 2015 μπορείτε να μας διασφαλίσετε, μπορείτε να μας πείσετε για την ικανότητά σας να είστε οι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Πεστε μας έναν ρεαλιστικό σας στόχο και πώς θα τον επιτύχετε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντική πρόκληση, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Είπα σήμερα ήδη ότι είναι απαραίτητο το αργότερο δε στο Παρίσι το 2015 να θεσπίσουμε κοινού δεσμευτικούς στόχους που θα ισχύουν όχι μόνο βεβαίως για την Ευρώπη. Μπορώ να σας πω ότι θα πράξουμε και στο Παρίσι κάθε τι που βρίσκεται μέσα στις δυνάμεις μας. Δεν έχουμε ακόμα συντονισμένο στόχο, δεν έχουμε ακόμα ορίσει κοινό στόχο, γι' αυτό δεν μπορώ να πω τίποτε για τα συγκεκριμένα νούμερα που θα ζητήσουμε να ισχύσουν και βεβαίως αφού οι εταίροι μας και ιδίω οι ΗΠΑ και η Κίνα πρέπει και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες των. Μπορούμε μόνο να πούμε ότι το περιβάλλον μας πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα, να μην επιδεινωθεί δηλαδή. Είμαι πεπισμένη ότι και οι άλλες χώρες γνωρίζουν ότι η στόχη αυτή είναι σημαντική. Χαίρομαι που οι μηχανισμοί αγοράς που διαθέτουμε στην Ευρώπη, όπως το σύστημα ETS, ε, εμπορίας των ε, δικαιωμάτων εκπομπών, έχει αποδείξει την αξία του. Και ο μηχανισμός αυτός γίνεται τώρα ενδιαφέρον και για την Κίνα. Είμαστε ήδη σε επαφές με την Κίνα και γι' αυτό έχω την ελπίδα ότι και άλλες χώρες θα υιοθετήσουν τους στόχους αυτούς. Ο κύριος Ρόιλ του Λαϊκού Κόμματος. Κυρία Υποψηφία Επίτροπε, θέσαμε πολλές ερωτήσεις για την Ενεργειακή Ένωση, παρόμοιες ερωτήσεις, δώσατε παρόμοιες απαντήσεις, δεν με εκπλήσει αυτό. Βέβαια υπήρξαν και κάποιες αμφιβολίες για την προηγούμενη πολιτική σας ζωή και εκεί δώσατε κάποιε απαντήσει. Είπατε τώρα ότι η Ευρώπη οφείλει να ομιλεί με μια φωνή και προ τα έσω, προ τι χώρες μέλη δηλαδή, αλλά και προ τα έξω, για παράδειγμα προ του ρώσου κτλ. Το ερώτημα τώρα είναι γιατί θεωρείτε ότι εσεί με τι δικέ σα προδιαγραφέ είστε ικανοί να τα υλοποιήσετε αυτά. Ποιε είναι οι δικέ σα ιδιαίτερε ιδιότητε, ποιε είναι οι ποιότητέ σα που θα επιτρέψουν να υλοποιήσετε αυτή την υπόσχεση. το ότι δώσατε παρόμοιες απαντήσεις σε παρόμοιες ερωτήσεις, για μένα αυτό είναι υπέρ σας, διότι δείχνει ότι έχετε μία γραμμή. Αλλά δώστε μου μια απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη Ευρωβουλευτή, αν θέλουμε να είμαστε ισχυρότεροι, πρέπει να έχουμε ένα κοινό μέτωπο έναντι των τρίτων χωρών, των εταίρων μας. Μπορώ να σας πω ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο όταν χρειάστηκε να δώσω μάχη και να πείσω τις χρηματοπιστωτικές αγορές διεθνώς ότι η Σλοβενία δεν θα χρεοκοπήσει, παρά το γεγονός ότι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτική εντός της Σλοβενίας αλλά και στο εξωτερικό ήταν απόλυτα πεπισμένοι ότι η Σλοβενία ήταν στο χείλος της καταστροφής. Με συγκεκριμένα μέτρα απέδειξα ότι δεν ε, στέκομαι μόνο στα λόγια, αλλά περνάω και στην πράξη. Και αυτό θα κάνω και ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν φυσικά μου δώσετε το χρήσμα και μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα. Βεβαίως και δεν είμαι μόνη μου. Οι συνάδελφοι επίτροποι και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αν χρειαστεί, θα συνεισφέρουν και αυτοί και θα ε, εργαστούμε με συνεκτικό ε, τρόπο και σε πνεύμα συνεργασίας. Τώρα, πέραν του ποιο θα είναι ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ε, θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό να μιλά όλο το σώμα των επιτρόπων με μία φωνή και να αποφεύγει ε, αποκλήσει μεταξύ των επιτρόπων. Και νομίζω ότι η νέα σύνθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η νέα τη δομή, όπω την προτείνει ο πρόεδρο Γιούνκερ, θα μα εγγυηθεί αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι ε, βέβαιη ότι η πείρα η οποία αποκόμισα τον τελευταίο 1,5 χρόνο που ηγήθηκα της ε, κυβέρνησης της Σλοβονίας στη χειρότερη στιγμή ε, στην ιστορία μιας τόσο νέας χώρας όσο η Σλοβενία θα με βοηθήσουν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Μπός. Ευχαριστώ. Κύριε Μπράτουσεκ, ε, ήσασταν είχατε θέση στη χώρα σας και μετά παραιτηθήκατε. Γιατί παραιτηθήκατε. Πιστεύω ότι θα, έπρεπε να είχατε συνεχίσει με τα καθήκοντά σας. Δεν είχατε λόγο να παραιτηθείτε. Και αν το είχατε κάνει, θα είχαμε άλλο υποψήφιο από τη θα είχε προταθεί άλλος υποψήφιο από τη Σλοβενία. Είναι ενδιαφέρον ότι στην αρχή δεν ήσασταν στον κατάλογο των υποψηφίων κατόπιν προβληθήκατε ως μοναδική υποψήφια. Αυτό δεν το θεωρώ πλώς ανήθικο, αλλά το θεωρώ διαφθορά. Και η Επιτροπή κατά τη διαφθοράς μελετά την υπόθεση. Τώρα το ερώτημα είναι, τι θα συμβεί αν από το αποτέλεσμα της έρευνας φανεί ότι δεν τηρήθηκε η νομοθεσία. Θα παρατηθείτε ή θα διατηρήσετε τη θέση σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά μου δίνετε την ευκαιρία να σας εξηγήσω τι συνέβη στη Σλοβενία όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Είμαι πεπισμένη ότι πρόκειται για εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι. Η Σλοβενία έστειλε ένα κατάλογο με τρεις υποψηφίους στις Βρυξέλλες. Δεν γνωρίζω τι είδους κατάλογο έχετε εσείς κατά νου, είδατε εσείς, αλλά ο μοναδικός κατάλογος που έστειλε η κυβέρνηση της Σλοβενίας προς τις Βρυξέλλες περιελάμβανε και το όνομά μου. Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ αποφάσισε, είχε τη δυνατότητα να επιλέξει κάποιον άλλο από τον κατάλογο. Υπήρχε και άνδρας και άλλη γυναίκα υποψήφιος. Αυτά όσον αφορά την επιλογή. Τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά μέχρι στιγμής στη Σλοβενία δεν είχαμε πρόβλημα. Δεν ήταν πρόβλημα. Εάν υπήρχε, ήσουν υποψήφιος για μία πολιτική θέση, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσες άλλη. Τα εσωτερικά πολιτικά θέματα στη Σλοβενία ξέφυγαν με τον τρόπο που έγινε, αλλά και προηγουμένως είπα ότι ποτέ ποτέ. Δεν είχα προβλήματα με το νόμο. Πρέπει να με πιστέψετε. Είμαι προσιλωμένη στον αγώνα κατά της διαφθοράς και η αστυνομία που ε, δύο και τη διαφθορά αλλά και το δικαστικό σύστημα λειτουργούσαν πλήρως όσο ήμουν Πρωθυπουργό. Ευχαριστώ κυρία Κέστιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακόμα δεν έχετε απαντήσει στην ερώτηση του προηγουμένου βουλευτού, δηλαδή αν θα παρετηθείτε εφόσον επιβεβαιωθούν οι υποψίες διαφθοράς ή εάν απαγγελθούν κατηγορίες λόγω διαφθοράς. Παρακαλώ πέστε μας καθαρά ναι ή όχι. Δεύτερη ερώτηση. Κρατικές εγγύησεις που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επίπεδο των 70 δισεκατομμυρίων λιρών για την έγερση νέου πυρηνικού εργοστασίου, καθώς και για 35 χρόνια εγγύηση ότι θα δύναται να παρέχει ρεύμα. Αυτά αντιτίθεται στη στήριξη στους νόμους περιστήριξης. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε αυτές τις σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Και ναι βέβαια το ενεργειακό μίξ είναι υπόθεση των χωρών μελών, εδώ όμως πρόκειται για αθέμητες επιδοτήσεις. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε ξεκάθαρα χωρίς να υπεκφύγετε. Ευχαριστώ. Απάντησα ήδη ότι γνωρίζω τι στάση πρέπει να τηρήσει ένας πολιτικός εφόσον έρθει σε σύγκρουση με τον νόμο. Ωστόσο, πέραν αυτού, θεωρώ σημαντικό να τονίσω και πάλι ότι στην προκείμενη περίπτωση καμία αρχή δεν έχει διαπιστώσει ότι πρόκειται περί διαφθοράς. Όταν εμφανίστηκα εντόπιον της Επιτροπής κατά της διαφθοράς, με διαβεβαίωσε ο ίδιος ο πρόεδρός της ότι εναντίον μου δεν υπάρχει απολύτως καμία δίωξη. Αυτό είναι το ένα θέμα. Τα πυρηνικά εργοστάσια τώρα. σας εξήγησα ποια είναι κατά τη γνώμη μου τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως όλες οι κρατικές επιδοτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους υφιστάμενους κανόνες. Κρατικές επιδοτήσεις δεν μπορούν να παραβιάζουν το δίκαιο. Όσον αφορά συγκεκριμένα τώρα Τα 27 δισεκατομμύρια για τα οποία μιλήσατε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θα πρέπει πρώτα να ενημερωθώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Αντιπρόεδρε Επιτροπέ, θα ήθελα κάποιες συγκεκριμένε ε, απαντήσεις και θα επικεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο ε, ζήτημα. Ε, χώρες, μέλη οι οποίες είναι απομονεμένες ενεργειακά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα συμπεράσματά της του 2011 και τα υπόλοιπα είπε ότι από το 2015 και τούδε δεν θα πρέπει κανένα κράτος μέλος να είναι απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Πόρο απέχουμε από αυτό. Ποια είναι το όραμά σα λοιπόν για τι χώρε μέλη οι οποίες είναι απόλυτα απομονωμένε από πλευρά ενέργειας και τι θα κάνετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι θα επιτευχθεί ε, ο στόχος αυτός. Υπάρχει συμφωνία της Μάλτας για την ε, κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου, αλλά χρειάζεται υποστήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδότηση. Τι θα κάνετε για να ε, εφαρμοστούν τα προγράμματα αυτά το συντομότερο δυνατόν. Και επίσης υπάρχει και ο κανονισμός TNI, ο οποίος υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν συγκεκριμένους κανόνες, πώς θα διασφαλίσετε ότι θα εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ja, e, pravzaprav se danes... Ne. Σήμερα μιλήσαμε αρκετές φορές ε, για τα προγράμματα υποδομών και γνωρίζω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δύο προβλήματα πρωτίστως. Οι χώρες νήσι, στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς, Και εδώ θεωρώ ότι έχουμε χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες και μετά από το 2009 ε, στη στρατηγική για την ασφάλεια εφοδιασμού αναφέρονται 33 προγράμματα τα οποία θεωρούνται κατεπήγοντα προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις υποδομές μας. Και αυτό βεβαίως αφορά και ε, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε εσείς. Αυτό λοιπόν είναι καθήκον μας και αυτή τη δέσμευση αναλαμβάνουμε. Αλλά τα προγράμματα τα οποία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί ή δεν έχουν ξεκινήσει, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το οποίο συνέβη στο παρελθόν. Τα προγράμματα βρίσκονται στο στάδιο στο οποίο βρίσκονται ή δεν έχουν καν ξεκινήσει και θα μπορούσα να σας πω ότι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου τα προγράμματα προτεραιότητας, τα οποία είναι πήγοντα και τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά ε, εντός ε, της στρατηγικής ε, για την ασφάλεια εφοδιασμού, θα πρέπει να υλοποιηθούν. γνωρίζω ότι η ενεργειακή ασφάλεια εξαρτάται ακριβώς από την εσωτερική αγορά και την ολοκλήρωσή της. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στην συνάδελφο κυρία Σπυράκη. Thank you, Chairman. Allow me to explain that uh, I insist to this question. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να επιμείνω γιατί εδώ, εδώ είμαι. Είναι θέμα αρχής για μένα κυρία υποψήφια Πρόεδρε, Στη διάρκεια των ε, εκλογών του 2014 στην ε, Σλοβενία, η εκστρατεία σας ήταν γεμάτη αντιευρωπαϊκά συνθήματα. Είπατε ότι σώσατε τη Σλοβενία από την Βρυξέλλες και τώρα ήρθατε εδώ να μας πείτε ότι σώσατε την Ευρώπη από το πρόβλημα της Σλοβενίας. Έχετε το δικαίωμα να αλλάζετε, αλλά το Viva Comunista δεν είναι αντιφασιστικό σύνθημα. Θεωρώ ότι είναι σύνθημα κατά των αξιών της Ευρώπης. Επιπλέον συμμετείχατε σε ένα αντιευρωπαϊκό, σε μια αντιευρωπαϊκή εκδήλωση. Είναι και αυτό αντιφασιστικό τραγούδι. Υπάρχει το ερώτημα πιστεύετε πραγματικά ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη θέση και από την άλλη και επιμένω από αυτού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας πιστεύω συμβιβάζονται με το ρόλο σας του Αντιπροέδρου. Σας ευχαριστώ. Γεια. Ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να απαντήσω για μία ακόμα φορά στο, για το ίδιο ζήτημα. Πρώτον, αυτά που λέμε πρέπει να είναι τεκμηριωμένα. Ποτέ δεν έγραψα ή ποτέ δεν, και ποτέ δεν είπα οτιδήποτε θα μπορούσα να με κάνει να εμφανιστώ ως αντιευρωπαία. Χαίρομαι, είμαι περήφανη που είμαι Σλοβένα, είμαι περήφανη που είμαι Ευρωπαία και είμαι πολύ περήφανη που ως Πρωθυπουργό κατάφερα να βγάλω τη χώρα μου από μια πολύ βαθιά κρίση χωρίς βοήθεια. Η Ευρώπη πρέπει να αισθάνεται περήφανη που η Σλοβενία έλυσε μόνη της τα προβλήματά της. Γιατί τελικά η επίλυση των προβλημάτων σε άλλων χωρών έχει στοιχήσει σε όλους τους Ευρωπαίους. Και γι' αυτό με υπερηφάνεια μπορώ να πω ότι αυτό που κάναμε εμείς το τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, αλλά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Επανήλθατε και πάλι στην εκδήλωση στην οποία συμμετείχα, στην οποία παραβρέθηκα. Ήταν μια εκδήλωση μνήμης ένας εορτασμός της εθνικής επαιτίου. Όλη η πολιτική ελίτ ήταν παρούσα. Προηγουμένως είπα ότι τραγούδισα ένα τραγούδι που στη Σλοβενία θεωρείται αντιφασιστικό. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι η Ευρώπη στηρίζεται σε κοινέ αξίες και άρα δεν χρειάζεται να απολογηθώ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κόφοντ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπράτσεκ. Εδώ είμαι. Σας έχουν αναθέσει ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο και πραγματικά προσπαθώ να αντιληφθώ τι θα κάνετε αν γίνετε επίτροπο. Στην αποστολή σας αναφέρετε σαφώς ότι πρέπει να εργαστείτε υπέρ της Ευρώπης ώστε να γίνει ο υπαριθμόν ένα παράγον στην, ε, ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μας έχετε δώσει ούτε μία ένδειξη όμως σήμερα του πώς ακριβώς θα επιτύχετε αυτό το στόχο. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να ακούσω από εσά αν έχετε κάτι κατά νου. Λέτε ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχει κάτι στο μυαλό σας το οποίο ε, θα μας μειώσει την ανταγωνιστικότητα εάν ε, πετύχουμε τους στόχους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μήπως ε, δεν είναι αρκετά φιλόδοξος ο στόχος που έχουμε για το 2020 και θα πρέπει να έχουμε καλύτερους στόχους. Και υπάρχει κάτι στην Ευρώπη ώστε να μπορούμε να εξάγουμε αποτελεσματικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, από τη μία χώρα στην άλλη. Πώς σκοπεύετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να το πιάσουμε από το τέλος. Επενδύσεις, επενδύσεις και ξανά επενδύσεις. θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσω ότι μεγάλο τμήμα των ε, χρημάτων που ανακοίνωσε ο κύριος Γιούνκερ θα αφορά επενδύσεις και προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας με επενδύσεις σε προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας επιτυγχάνουμε δύο στόχους. Μειώνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ταυτόχρονα επιτυγχάνουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους, τους στόχους της κλιματικής αλλαγής και δεύτερον μειώνουμε την εξάρτησή μας από εισαγωγές. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη θα γίνει πιο ανεξάρτητη ενεργειακά. Οι στόχοι. Όπως ε, επανέλαβα σήμερα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι στόχοι πρέπει ακόμα να συμφωνηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η διάθεση είναι μέχρι το 2030 να εγγυηθούμε 27% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, στο ενεργειακό μείγμα. Αυτός ο στόχος για κάποιες χώρες μέλη μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα, ενώ για κάποιες άλλες είναι πιο δύσκολος. Και παρά το γεγονός ότι σήμερα επανέλαβα το ίδιο, ε, τα κράτη-μέλη βάσει της συνθήκης είναι ανεξάρτητα και υπεύθυνα μόνα τους για ο καθορισμό του ενεργειακού του μείγματος. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συνθήκη, να παραβιάσουμε τη συνθήκη. Αυτοί είναι οι κανόνες και αν έχουμε ένα στόχο και είναι κοινός αυτός ο στόχος, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα επιτυχής αποτέλεσμα. Και τώρα ο συνάδελφος Νούνο Μέλιο. Comissário nomeada, a dependência energética Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης μπορεί να φτάσει στο 80% μέχρι το 2025. Αυτός ο βαθμός εξάρτησης θα πρέπει να αντιστραφεί. Άκουσα σήμερα ότι η Πορτογαλία και η Ιβηρική Χερσόνησος μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στον χώρο αυτό. Έχουμε από τα 11, 11 ε, σταθμούς φυσικού αερίου στην Ευρώπη και μπορούμε να αντικαταστήσουμε το 57% των ε, εισαγωγών της Ευρώπης από τη Ρωσία αν τα δίκτυα λειτουργούν. Όμως μόνο το 1,6% ε, υπάρχει στην Ιβηρική σχερσόνικα. Το Συμβούλιο της Βαρκελόνης του 2002 έθεσε ένα στόχο 10% μέχρι το 2012 θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τη Ρωσία μέσω Πορτογαλίας και Ισπανίας αν υπήρχαν αυτά τα δίκτυα. Μπορείτε να μου απαντήσετε συγκεκριμένα λοιπόν ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βουλευτή για το ερώτημα αυτό. Για μία ακόμα φορά θα επανέλθω στο θέμα των υποδομών. οι υποδομές είναι ο λόγος για τον οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί η εσωτερική μας αγορά. Επανειλημμένως υπογραμμίζω ότι πρέπει να συνδεθούν τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες και η κάθε περιοχή εντός των κρατών μελών, ώστε να εξασφαλιστεί η μεταφορά της ενέργειας. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας με όσα είπατε. Απλώς για μία ακόμα φορά πρέπει να επαναλάβω ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να δημιουργηθούν οι τόσο απαραίτητες υποδομές το ταχύτερο δυνατόν. Δεν μπορώ από μόνη μου να αλλάξω τα πράγματα. Κυρίως πράγματα που θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει υπήρξαν ευκαιρίες που χάθηκαν. Όμως πρέπει να αρχίσουμε τη δουλειά, πρέπει να προχωρήσουμε πρόσω ολοταχώς και σαφώς ο πρόεδρος Γιούνκερ ανέφερε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του πακέτου θα κατευθυνθεί προς τις υποδομές ενέργειας. Μόνο μια διασυνδεδεμένη εσωτερική αγορά μπορεί να εξασφαλίσει ε, μια καλά λειτουργούσα και ανθεκτική ενεργειακή νότα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρότε. Ο κύριος Γκρότε, ως μελλοντική υποψήφια αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, Επιτροπής δεν μιλήσατε για τις εκπομπές αερίων ούτε μία φορά για σας. Ποια είναι αποδεκτή τιμή για τον τόνο του διοξιδίου του άνθρακος. Θα υποστηρίξετε τη σταθερότητα των αγορών. Πόσα πιστοποιητικά διοξιδίου του άνθρακος πρέπει να απομακρυνθούν από το εμπόριο πιστοποιητικών έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το εμπόριο να λειτουργήσει πραγματικά, να αποδώσει πραγματικά. Η υποψήφια επιτροπός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευρωβουλευτά για την ερώτησή σας. Ίσως ήταν πράγματι λάθος μου που δεν το ανέφερα αυτό. Βέβαια κανείς από εσάς δεν ρώτησε κιόλας. Να σας πω ωστόσο λίγα λόγια σχετικά. Πιστεύω ότι ο μηχανισμός αυτός χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικός για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουμε θέσει. Είναι δύσκολο να καθορίσουμε την τιμή. Την τιμή θα την καθορίσει η αγορά. Είναι γεγονός ότι η κρίση, ας το πω έτσι, η κρίση άφησε τέχνη της και σε αυτό τον τομέα. Και η τιμή είναι σήμερα χαμηλότερη, του τόνου δηλαδή, του διοξιδίου του άνθρακος από ό,τι θα αναμέναμε. Υπάρχει πρόταση να εισαχθούν αυτά τα αποθεματικά στην αγορά ώστε να αφαιρεθούν πιστοποιητικά από το, τα στο εμπόριο μέχρι το 2021. Εγώ πιστεύω ότι ο μηχανισμός αυτός είναι σημαντικός. και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια ώστε να λειτουργήσει το σύστημα αυτό και στο μέλλον. Πιστεύω ότι με τον μηχανισμό αυτό θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους, που είναι πράγματι πολύ σημαντικοί. Υποστηρίζω εν τέλει την εισαγωγή αυτού του σταθεροποιητικού της αγοράς μηχανισμού. Ε, ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση, ο κύριος Λίζε από το Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία υποψήφια Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια ευκαιρία ακόμη να απαντήσετε συγκεκριμένα. Δεν έχουμε μόνο τα δύο λεπτά της απαντήσεώς σας, μπορείτε να απαντήσετε και στα πέντε λεπτά της καταληκτικής σας ε, τοποθέτησης. Πρώτον, ο εταίρος σας, Αρίας Κανιέτε, ανέλαβε την Τετάρτη πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Είπε 30% αποδοτικότητα της ενέργειας ως δεσμευτικό στόχο. Αύξηση των επενδύσεων. Είπε ότι είναι διατεθειμένος να προτάξει μάλιστα τον μηχανισμό αυτό. Μίλησε και για τους στόχους μετά το 2030 και μάλιστα μίλησε με συγκεκριμένα λόγια. Γνωρίζετε τις δεσμεύσεις αυτές που ανέλαβε ο Αρίας Κανιέτε. Θα τον υποστηρίξετε ή εν αμφιβολία θα τον σταματήσετε, θα ανακόψετε την πορεία του. Τέλος είπα το τραγούδι εκείνο είναι αντιφασιστικό και αναφέρεται ωστόσο στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να κατανοήσετε ωστόσο ότι αυτό κάπως έχει προκαλέσει ανησυχίες μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, Ευχαριστώ ε, κύριε Ευρωβουλευτά. Το τραγούδι. Νομίζω το εξήγησα. Ας ξαναπώ μια φορά. Στη Σλοβενία το τραγούδι έχει χαρακτήρα αντιφασιστικό. Το τραγουδούσαν και άνθρωποι όταν έριξαν το καθεστώ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δεσμεύσει του κ. Κανιέτε, τις γνωρίζω. Είπα λοιπόν σήμερα κατά επανάληψη ότι έχουμε πρόταση τώρα κατατεθειμένη που λέει τουλάχιστον 27% φορείς ανανεώσιμης ενέργειας, 30% απόδοση της ενέργειας, αποδοτικότητα της ενέργειας. Και εγώ ίδια υποστηρίζω τους στόχους αυτούς. Πάει να πει ότι οι συνάδελφοί μου και εγώ συμφωνούμε. Και όπως προανέφερα, πιο σημαντικό και από τον καταμερισμό των ευθυνών, των αρμοδιοτήτων, ακόμα πιο σημαντικό είναι όλοι να μιλούμε με μια φωνή και όλοι να αγωνιζόμαστε υπέρ κοινών στόχων. Αυτό το τονίζω και πάλι. Κοινός μας στόχος θα είναι για το έτος 2050 και νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό και θα χρειαστεί να συμφωνήσουμε και με άλλες χώρες εταίρους. Λοιπόν, στόχος μας πρέπει να είναι να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 80% μέχρι το 2050. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συμφωνήσουμε και με τους άλλους εταίρους μας και να συμφωνήσουμε πάνω σε κοινούς στόχους και αυτό θα επιδιώξω. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω επισήμως όλους τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους και την υποψήφια επίτροπο για τις απαντήσεις της. Είναι σαφές ότι Ίσως όλοι οι συνάδελφοι περίμεναν κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες, γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να καλέσω την υποψήφια επίτροπο να κάνει την ε, ε, τελική της δήλωση. Έχει πέντε λεπτά ε, στα οποία θα έχει τη δυνατότητα να μας δώσει κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες και λεπτομέρειες τις οποίες ίσως δεν μπόρεσε να συμπεριλάβει στο χρόνο που είχε για να δώσει απαντήσεις. Ο λόγος στην Επίτροπο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις και για το γεγονός ότι μου δώσετε τη δυνατότητα να απαντήσω. Ευχαριστώ και τον κύριο Γιούγκερ που μου έδωσε τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια παραπάνω για το όραμα της ε, Ενεργειακής Ένωσης και να σας δώσω και κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση η οποία επιβάλλει ε, να αναλάβουμε δράση. Μετά το 2009 δεν έγιναν αρκετά για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού. Πρέπει να έχουμε μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με το βλέμμα στο μέλλον. Και οι στόχοι δηλαδή μια ε, κλιματική πολιτική με το βλέμμα στο μέλλον είναι σαφής. Κυρίως οι στόχοι του 2020. 20% μείωση των ε, αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου, 20% ε, ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 20% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. η στόχοι αυτή θα έχουν συνέχεια τους στόχους για το 2030. 30% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να υλοποιήσουμε προγράμματα μείωσης τη ενεργειακή κατανάλωση που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε την περιβόητη πράσινη οικονομική ανάπτυξη. Και επίσης 27% ε, τουλάχιστον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ο στόχος ο οποίος ανέφερα και προηγουμένως για το 2050 και θεωρώ ότι θα έχουμε και υποστήριξη από τις πόλπες χώρες εταίρους, επ' αυτού είναι η μείωση κατά 80% των εκπομπών. Τα βασικά στοιχεία της Ενεργειακής Ένωσης στοιχεία τα οποία προέκυψαν και από την σημερινή συζήτηση είναι καταρχάς καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε καλύτερες υποδομές, καλύτερη διασύνδεση, μια ε, πιο ισχυρή οικονομική αγορά που θα μας επιτρέψει να δώσουμε κίνητρα για ανταγωνιστικότητα που είναι πολύ σημαντική και για την ε, βιομηχανία αλλά και για τους πολίτες. Στο παρελθόν είχαμε μια οικονομία υψηλή κατανάλωση άνθρακα. Το πέρασμα στην οικονομία χαμηλή κατανάλωση άνθρακα θα μπορέσουμε να το κάνουμε ε, μέσω ε, ενεργειακής αποδοτικότητας και μέσω αυτών των στόχων θα καταφέρουμε να μειώσουμε και την εξάρτηση από τις εισαγωγές. Και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινή μας δράση ενώπιον των διεθνών μας εταίρων. Όσο μεγαλύτερη βαρύτητα όσο μεγαλύτερη ισχύ ε, έχουμε τόσο καλύτερο. Και αυτό φυσικά θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε εάν μπορούμε να δράσουμε από κοινού και αν μπορούμε να διασφαλίσουμε και μία κοινή θέση. Αυτό το οποίο αποτελεί για μένα προτεραιότητα, εάν μου δώσετε το χρήσμα, θα ε, είναι να καθορίσω με τους συνεργάτες μου ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. ένα σχέδιο για το μέλλον, για το ενδεχόμενο έλλειψης φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Οι συνεργάτες μου ήδη ετοιμάζουν το σχετικό έγγραφο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο ε, προσεχώς και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι υπάρχει όραμα, υπάρχουν οι στόχοι και έχουμε ξεκινήσει μία άγουσα η οποία θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ κυρία Αλένκα Μπράτουσεκ, υποψήφια αντιπρόεδρε και επίτροπε. Ευχαριστούμε για την καταληκτική αυτή δήλωση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από τις δύο επιτροπές, όπως επίσης και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής κοινή Γνώμης, είτε όσους παρίστανται, αλλά και αυτούς που μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου. Θα ήθελα να σας δώσω τελικές πληροφορίες για την Επιτροπή Ήτρε. Σήμερα το βράδυ στις 8 θα γίνει συνεδρίαση συντονιστών, ενώ αύριο όλοι μας όλα τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Έχουμε την ακρόαση του κυρίου Γιούρκη Κατάινεν στις 10 το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τους συναδέλφους της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Η συνεδρίασή μας για την εξιολόγηση θα γίνει από τις 7.30 έως τις 9 σήμερα το βράδυ με τους συντονιστές και κατόπιν θα ξεκινήσει η κοινή συνεδρίαση ε, συντονιστών επιτροπών Ήτρε και Ένβη από τις 9 ως τις 10. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.